Um, μπορούμε να καθίσουμε σας παρακαλώ για να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα στην ημερήσια διάταξη και μόλις άκουσα ότι ο πρόεδρος μας κύριος Λόπες το έχει καθυστερήσει λίγο. Θα έρθει λίγο αργότερα λοιπόν. Πρότεινα όμως να ξεκινήσουμε. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν είμαι 100% προετοιμασμένη για τις συνεδρίες, θα κάνω όμως ό,τι μπορώ. Έχουμε αρκετέ ψηφοφορίες, θα προσπαθήσω να τις προχωρήσω δυνατόν πιο γρήγορα. Και πριν ξεκινήσουμε, θα μου επιτρέψετε να σας επισημάνω τα εξή δύο τις δύο εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πρόσφατα γεγονότα και τι εξελίξει στην Ισία, την Αίγυπτο, τη Λιβύα και άλλε χώρε. Θα συζητηθούν λοιπόν αυτέ οι εξελίξει σήμερα στην Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων από τι 6.30 έω 8 και κλεισμένων των θυρών, την παρουσία και του Επιτρόπου Φιούλε και του πρεσβευτού Δήμου, και δεν μα λέει πού είναι πρέσβη αυτό. και αύριο το πρωί στην Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών από τις 9 και μισή παρουσία της, της του Συμβουλίου, της Επιτρόπου Μάλστρομ και του Διευθυντού της Frontex κυρίου Λάτινεν. Αν λοιπόν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις προς την ημερήσια διάταξη, παρακαλώ να την εγκρίνουμε. Περνάμε απευθεία στις ε, ψηφοφορίες. Έχετε φέρει όλες τις κάρτες σας για την ψηφοφορία. Πρώτη ψηφοφορία πρόκειται για την έκθεση του κυρίου Φαντανικάπου ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους. Ξεκινούμε λοιπόν την ψηφοφορία. Τροπολογία περιθμών 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Νομίζω δεν ψηφίζουν οι αντιπρόεδροι. Θα πρέπει να ενωθείτε με τον όχλο αν θέλετε να ψηφίσετε. Δεύτερη ψηφοφορία. Τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρία σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται και αυτό. Ας επαληθεύσουμε το δεύτερο τμήμα λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τις ψηφοφορίες. είναι υπερβολικά πολύ φιλελεύθεροι, αλλά δεν νομίζω ότι έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν μπορεί ποτέ να περισσεύουν φιλελεύθεροι στον κόσμο μας. Λοιπόν, ας φύγει ένας. Να είμαστε εντάξει με τα νούμερα. Είκοσι υπέρ, άρα εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Α, έχουμε και τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές το πιστεύω επαληθεύουμε άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι εγκρίνεται Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, Τέσσερα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται βλέπω αλλά Ας επαληθεύσουμε την 7 άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε παρακαλώ. Μάλλον έχει απορριφθεί, αλλά σε επαληθεύσουμε τη 10, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρασε τη ψηφοφορία. Όντω απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές μάλλον απορρίπτεται, αλλά ας το επαληθεύσουμε την 12 τροπολογία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρας. Απορρίπτεται όντως. Ίσα ίσα, 13 υπέρ, κατά αποχές 13 λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. πέρα. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Θέλετε να επαληθεύσουμε τη 14. 14 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές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 Σάιμον, ναι. Ωραία. Πέρας προφορές λοιπόν, αφού ψήφισες και εσύ. Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική είχατε Καλός καλώς ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας εγκρίνεται με ευρύτατη πλειοψηφία. Προχωρώ στην επόμενη ψηφοφορία και τον επόμενο κατάλογο. Το επόμενο θέμα είναι η μετανάστευση. Πρόεδρε, διαδικαστικό. Πρόεδρε, δεν μας είπατε το αποτέλεσμα της πληροφορίας. Δεν το δείξατε. Δεν το δείξε η οθόνη. 30 υπέρ και 5 κατά χωρίς κάποια εποχή. Ζητώ συγγνώμη, είχα την ότι αυτά που βλέπω εγώ στη μικρή μου οθόνη τα δείχνει και η μεγάλη της αίθουσας, αλλά φαίνεται ότι ε, έχω προνομιακή πρόσβαση σε πληροφορίες. Επόμενο θέμα λοιπόν, έκθεση Κέλλερ ως προς τις ε, μεταναστευτικές ροές που προκύπτουν λόγω της αστάθειας, πεδίο και ρόλος ευρωπαϊκής πολιτικής, ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Θέλετε σε τμήματα ψηφορία κυρία Χολμάιερ. Θέλετε να το ζητήσετε τώρα, πριν από την έναρξη ψηφορία, παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω στη συμβαστική πρόταση 4 ε, σε τμήματα, μέχρι το displacement ένα τμήμα και μετά ένα δεύτερο από το σημείο ζητή από την Επιτροπή Ask the Commission μέχρι το ε, μακροπρόθεσμες λύσεις, εξέβρεση μακροπρόθεσμων λύσεων. Το έχετε όλο το κείμενο. Η Πρόεδρος, νομίζω ότι η ποιότητα του ήχου είναι πολύ κακή σε αυτήν την αίθουσα. Ε. Αν μπορούν οι τεχνικοί να μας βοηθήσουν, υπάρχει αντι... Ε, αντίλαλος εδώ. Ο κύριος μπορεί να αποσύρει όταν έρθει η ώρα την τροπολογία του. Ξεκινώ λοιπόν την ψηφοφορία με την συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και έτσι περνάμε στην 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θα έλεγα αλλά ας ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία 25, τροπολογία 25. Ψήφισαν όλοι. Ακόμη και αυτοί που άλλαξαν γνώμη μεταξύ μπορούμε να τελειώσουμε την ψηφοφορία εδώ. Καλώς. Απορρίπτεται. 27 τώρα, Χολμάιερ, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 4 το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε Δεύτερο τμήμα. Φαίνεται να είναι μισή-μιση η έκβαση της ψηφοφορίας. Δεύτερο τμήμα της συμβαστικής 4 παρακαλώ. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 19 υπέρ, 17 κατά. Τα βλέπετε τα αποτελέσματα άλλωστε. Φαίνεται ότι ψηφίζουν 9 από τους φιλελευθέρους αντί για 8. Εγώ βλέπω 8 λέει η κυρία Νότφελτ Μάλιστα. Σας βλέπω τώρα κύριε Γιούσεφ. Ένα ε, ένας από τους φιλελεύθερους πρέπει να σταματήσει να ψηφίζει. Ίσως εγώ. Και είναι και πιο καλή λύση νομίζω γιατί έτσι μπορώ να επικεντρωθώ στην καθοδήγηση προφορία. Α μην ψηφίσω εγώ λοιπόν. Α, να και ο πρόεδρο. Σοφή. Οχτώ ψήφου έχουμε. Έχουμε δικαίωμα για οχτώ ψήφου και είμαστε οχτώ στην αίθουσα. Όχι, είμαστε εννέα, είμαστε εννέα. Εννέα είναι τα μέλη των φιλελευθέρων. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, δεν θα σας είδα. Την άλλη φορά θα ζητάμε να φοράει καθένα το, το μπλουζάκι της ομάδα του για να αναγνωρίζουμε. Ναι, και ήρθε ο Πρόεδρος να αναλάβει εκείνος, παρακαλώ. Μόλις ψηφίσαμε τη συμβαστική 4. Αλλά είχαμε τον κύριο Μπουσετήλ. Ποιος στο λόγο. Τότε, Πρόεδρε, μια και ήταν υπεράριθμη η φιλελεύθερη, δεν θα έχει αλλάξει. 18-17 θα ήταν το αποτέλεσμα. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Μήπως να μην... Μήπως μια και ήταν άκυρη ψηφοφορία και μπορεί να ανατραπεί το αποτέλεσμα. Και έρχεται και ένα νέο μέρος από την ομάδα μου τώρα. Ε, ήταν άκυρη ψηφοφορία. Τι να κάνω εγώ. Δεν ξέρω αν μετά από αυτή την συζήτηση είδε κανείς το φως της αληθείας. Ας ξαναψηφίσουμε το δεύτερο ημίση τη συμβαστική 4, άρχεται η ψηφοφορία και εγώ δεν ψηφίζω. Δεύτερο ημίση τη συμβαστική 4. Ψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Μήπω περισσεύει κανένα σοσιαλιστής τώρα. <laughs> Ω, ενδιαφέρον το αποτέλεσμα. Δεν προσέχετε τι ζητάτε κύριε Μπουσούτιλ. Τι μπορεί να εκπληρωθεί. Um, Ευχαριστώ πολύ, Σόφη. Έρχομαι κατευθείαν από το αεροδρόμιο. Σας ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Αναλαμβάνω τώρα εγώ την Προεδρία και συνεχίζουμε με την τροπολογία 34. Υπέρ. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται, μάλλον αλλά σε επαληθεύσουμε. Πέρας. 20 υπέρ, 17 κατά, εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά. Αποχές. 37 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές σαν να είναι μοιρασμένο το αποτέλεσμα σε παληθεύσουμε άρχιτα φορεία. πέρας 21 ε, υπέρ, 17 κατά εγκρίνεται. 42 με προφορική τροπολογία τη εισηγήτρια. Όχι, ζητώ συγγνώμη, 40, 40, 40 είμαστε. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 41 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 42 τώρα με την προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ συμβαστική 5 σε τρία τμήματα μάλιστα σε, στο πρώτο τμήμα λοιπόν υπέρ κατά αποχές μάλλον εγκρίνεται θέλετε να επολυθεύσουμε ευχαριστώ το πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία Πέρα ψηφοφορίας να 22 υπέρ, 16 κατά. Δεύτερο τμήμα. Εγκρίθηκε λοιπόν. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Τώρα εγκρίθηκε. Και τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46. Κυρία Χολμάιερ. Η 46 νομίζουμε ότι έχει καλυφθεί από τη συμβαστική 5 και την αποσύρουμε. Με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος, δεν είχα προλάβει να προσαρμόσω τα ακουστικά μου. Σας ακούω τώρα. Πρόεδρε, νομίζουμε ότι το, η τροπολογία 46 καλύπτεται από τη συμβαστική 5 και άρα έχει καλυφθεί το θέμα. Αποσύρουμε λοιπόν την τροπολογία. Καλώς. Απεσύρθη 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές.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 κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά Αποχέ. απορρίπτεται 17 όχι, είχε απορριφθεί, ναι. Άρα την 17 όπως έχει προφορική τροπολογία από την είναι υπέρ κατά αποχές απορρίψετε 18 θέλετε παλήθευση σε 17 άρχεται η ψηφοφορία τη 17, πέρας προφορίας, 21 υπέρ, 16 κατά. Εγκρίνεται επομένω. 18 τώρα υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δύο τμήματα νομίζω ότι υπάρχουν στην 17. Είχαμε μια προφορική τροπολογία σε δύο τμήματα, έτσι δεν είναι. Πρόεδρος. Εγώ λέω πρώτα έχω αντιληφθεί ότι έπρεπε να ψηφιστεί προφορική, η τροπολογία 17 με την προφορική τροπολογία τη ηγήτρια, όπω έχει. Λάθο έχω καταλάβει. Κύριο Μπουσούτιλ, όχι γιατί θέλαμε να υπερψηφίσουμε με την τροπολογία, αλλά να κάτι τα ψηφίσουμε την προφορική. Θέλουμε να ψηφιστεί η προφορική τροπολογία. Αλλιώς δεν γίνεται δεκτή η υποβολή της τους ή άλλως. Μα εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε μαζί με την προφορική τροπολογία, έτσι Μα δεν φέρατε αντίρρηση στην υποβολή προφορικής τροπολογίας. Πρόεδρε, δεν ξάχαγατε την ψηφοφορία και εμείς νομίζαμε ότι ψηφίσαμε το πρώτο τμήμα. Και την υπερψηφίσαμε γιατί αυτό λέει το ο κατάλογος των ψηφοφοριών μα. Αλλά για την προφορική τροπολογία σκοπεύαμε να την καταψηφίσουμε. Πρόεδρος, εγώ δεν είδα να προβάλλει κανεί αντίρρηση. Μάλλον δεν, έχω λόγο να ε, μην ακολουθήσω αυτό που λέτε, αλλά, αλλά ε, είπα ότι ψηφίζουμε την τροπολογία με την προφορική τροπολογία τη συγκητρίας και δεν έφερε κανεί αντίρρηση. Κάνω λάθο. Κανείς δεν έφερε αντίρρηση. Κανείς δεν έφερε αντίρρηση στην ψηφοφορία με προφορική τροπολογία. Κυρία Ζόμερ, Πρόεδρε, αν κοιτάξετε λίγο στο κατάλογο, προβλέπονται δύο ψηφοφορίε στην τροπολογία 17. Μία χωρί την προφορική τροπολογία και μία με την προφορική τροπολογία. Εξού και εμείς ψηφίζουμε μόνο το πρώτο κομμάτι, χωρίς προφορική τροπολογία. Γιατί 17 προβλέπονται δύο χωριστές ψηφοφορίες, αναφέρονται στον κατάλογο. Παρακαλώ, κοιτάξτε το. Κυρία Κέλλερ, εσείς. Δεν ξέρω τι πρόβλημα έχει ο δικός σας ο κατάλογο Ο δικός μου όμως, που μου έχει αποστείλει γραμματεία ξεκάθαρα δείχνει ότι δεν είναι δύο χωρίς ψηφοφορίε, αλλά μόνο μία. Και προφορική τροπολογία. Και οι συστάσεις μου είναι είτε κατά χωρίς προφορική τροπολογία ή υπέρ με την προφορική τροπολογία. Δεν ξέρω πόσο ξεκάθαρο, πιο ξεκάθαρο θα μπορούσε να είναι στο κατάλογο των ψηφοφοριών αυτό. Μία ήταν η ψηφοφορία με την προφορική τροπολογία, κύριε Μπουσούτη. Τότε, πρόεδρε, θα πρέπει να αντιταχθώ στην υποβολή προφορικής τροπολογίας, δεν μπορεί να ψηφιστεί. Με συγχωρείτε, πρόεδρε. Όχι, ε, πρέπει να σεβαστεί το σκοπό μας ως προς την ψηφοφορία, την πρόθεσή μα, δηλαδή. Και εμείς θέλαμε να ψηφίσουμε όπως έχει το κείμενο. Όπως είπατε εσείς, Πρόεδρε, ακριβώς αυτή τη φράση χρησιμοποίησατε. Όπως έχει. Χωρίς δηλαδή προφορική τροπολογία. Κύριε Χολμάια, θα πρέπει να είναι δυνατόν, Πρόεδρε, ε, να επαναληφθεί μια ψηφοφορία για την οποία αμφισβητείτε το αποτέλεσμα της ψήφου. Αλλιώς τι δημοκρατία έχουμε και τι κοινοβουλευτισμό. Πρόεδρος, πολύ ευχαριστώ ε, να επαναλαβούμε την ψηφοφορία δεν μπορώ να ε, αποκλείσω ότι ενδεχομένως λόγω διαφορετικών εκδόσεων του κειμένου να έχει προκύψει κάποιο σφάλμα του καταλόγου του ψηφοφοριών. Εγώ έχω κατάλογο ψηφοφορία όπου βλέπω την ε, τροπολογία 17 της κυρία Τάνια Φαϊών τροποποιημένη με την προφορική τροπολογία της εισηγητρίας. Μπορούμε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Κλοντ. Ίσως πρόεδρε να διευκολύνουμε εάν αποσύρουμε την προφορική τροπολογία. Η Τάνια δεν είναι εδώ, αλλά την τροπολογία ολόκληρη, όχι την προφορική, την τροπολογία. Ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα απεσύρθη η προφορική τροπολογία και ψηφίζουμε την ε, βάση, τη βασική τροπολογία. Όχι, Θέλετε να την παραλάβουμε, κύριε Μπουσούτιλ. Πρόεδρε, είχε εγκριθεί χωρί προφορική τροπολογία. Και ξέρετε, εμεί είμαστε ευχαριστημένοι γιατί δεν θέλαμε την προφορική. Άρα έχει εγκριθεί χωρί την προφορική τροπολογία. Είναι σαφέ, κυρία Κέλλερ. Είτε δεχόμαστε ότι έγινε ψηφοφορία και άρα ψηφίσαμε μαζί με την προφορική και την εγκρίναμε, είτε δεν έχουμε ψηφίσει και ξαναψηφίζουμε χωριστά. Και οι σοσιαλδημοκράτε λένε ότι αποσύρουν ολόκληρη την τροπολογία και άρα δεν υπάρχει λόγο να την ψηφίσουμε. Εσεί θα το αποφασίσετε βέβαια. Είτε έχουμε όμω εγκρίνει όλο το κείμενο, είτε έχει αποσυρθεί η βασική τροπολογία από του σοσιαλδημοκράτε. Ο πρόεδρο. Ωραία. Θα γίνει από την αρχή όλη η ψηφοφορία και αυτό είναι ο πιο απλό τρόπο να επιληθεί το ζήτημα. Ψηφίζουμε τη 17 χωρί χωρίς προφορική τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η, τροπολο... η ψηφοφορία, η 17, χωρίς την, χωρίς την προφορική. Γιατί να μην τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Απλά τα πράγματα. Την έχουμε αποσύρει, Πρόεδρε. Πρόεδρε, είναι σφαλμένη η λύση στην οποία καταλήγεται και στις δύο περιπτώσεις. Είτε, όπως λένε οι συνάδελφοι, ήδη ψηφίσαμε και άρα απλώς μπερδεύτηκαν οι χριστιανοδημοκράτες και δεν ξέραν τι ψηφίζανε, είτε έχουν την ευκαιρία τους οι χριστιανοδημοκράτες, αλλά έχουν την ευκαιρία τους οι χριστιανοδημοκράτες και αποσύρουν την τροπολογία 17. Και εσείς ούτε τη μία λύση έχετε ακολουθήσει, ούτε την άλλη. Πρόεδρος έγινε μια ανακοίνωση ότι αποσύρεται η προφορική τροπολογία. Όλη η τροπολογία. Α, όλη η τροπολογία. Ναι, Πρόεδρε, οι σοσιαλιστές ζητούν την απόσυρση όλης της τροπολογίας. Άρα δεν υπάρχει λόγος σε ψηφοφορία για το θέμα αυτό. Όχι, καθόλου. Διαγράφεται ολόκληρη η τροπολογία. 18. 18 λοιπόν. Υπέρ. Then 19. Τη 19 τότε, εφόσον έχουμε ψηφίσει τη 18. Υπέρ. Υπέρ της 19. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20. Πάλι το ίδιο. Έχουμε μια προφορική τροπολογία ε, από την εισηγήτρια. Τη διατηρούμε ή όχι. Αποσύρεται η τροπολογία η προφορική ή όχι. Κλόντ, έχεις να πεις τίποτα για την τροπολογία 20. Παραμένει η τροπολογία 20, υπάρχει προφορική τροπολογία και απλώς λέει ο κατάλογος πληροφορία ότι η συγγήτρια υποφαινόμενη εμπροκειμένο Είμαι υπέρ ε, αν συμπεριληφθεί η προφορική τροπολογία και κατά αν όχι. Δηλαδή είναι μία ψηφοφορία συμπεριλαμβάνοντας και την προφορική τροπολογία. Κύριε Μπουσούτιλ. Εμείς διαφωνούμε με την προφορική τροπολογία, κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα. Αποσύρεται η προφορική τροπολογία, οπότε δεν υπάρχει λόγος να την ψηφίσουμε. Ωραία. Τροπολογία 21, υπέρ. Κατά. Εποχές. Ε, απορρίπτεται. Τώρα θα γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο τροποποιημένου κειμένου. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρα. Πέρας. Δεκαεννέα υπέρ, τρεις κατά, οπότε εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Yes, Mr. Μάλιστα, κύριε Καμάρε. Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια. Εγώ δεν διαφωνώ με, τη, το να αποσυρθεί ολόκληρη η τροπολογία 17. Θα ήθελα όμως να κατανοήσω το εξής. Γίνεται να ε, αποσύρουμε μια τροπολογία εφόσον έχει ψηφιστεί από την Επιτροπή. Ε, οι κανόνες το επιτρέπουν αυτό. Μπορεί αυτό να γίνει από οποιαδήποτε πολιτική ομάδα. Πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνω ότι έκαναν λάθος ε, στον κατάλογο ψηφοφορίας ε, οι ε, συνάδελφοι του ΕΛΚ. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά αν εγώ κάνω το ίδιο λάθο, ελπίζω να τύχω και εγώ τη ίδια ανοχή, γιατί δεν θα θέλα δύο διαφορετικού κανόνε να ισχύουν για τι μεγάλε και τι μικρέ πολιτικέ ομάδε. Απλώ ζητώ συζητώ αυτό το διαδικαστικό ζήτημα ε, μετά την ψηφοφορία, το θέτω. Γιατί εμείς κάποια στιγμή το είχαμε ζητήσει και δεν ήταν η ίδια μας η αντιμετώπιση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ε, εσείς ως πρόεδρος ε, δείχνετε μεγαλύτερη ανοχή στις μεγάλες ομάδες, μικρότερη ανοχή στις μεσαίες ομάδες και καμία ανοχή στις μικρές ομάδες πρέπει να δέχεστε το διαδικαστικό ε, αίτημα από όλες τις ομάδες ε, αδιακρίτως. First, Καταρχάς, να μας πει η νομική υπηρεσία σε σχέση με το νομικό υπόβαθρο της ερμηνείας ε, που έγινε με τη δυνατότητα, για τη δυνατότητα απόσυρσης μιας τροπολογίας όπως ε, πρότεινε ο συντονιστής ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών, που είναι και η ομάδα της οποίας μέλος ε, ε, πρότεινε το συγκεκριμένο κείμενο. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω το εξής. Προσπαθώ να σέβομαι εξίσου όλες τις πολιτικές ομάδες Επίσης προσπαθώ να χειριστώ καταστάσεις και ειδικότερα ε, δύσκολες, αντιφατικές καταστάσεις με... παραμένοντας λογικός. Προσπαθώ να ακούσω τις απόψεις όλων και προσπαθώ να καταλήξω σε μια συνενετική λύση αποδεκτή από όλους. Αυτός είναι ο δικός μου τρόπος. Ε, δεν βλέπω πώς γίνεται να δίνει κανείς μεγαλύτερο βάρος ή να ευνοεί τις μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες. Ή να έχει διακριτική συμπεριφορά κατά των μικρότερων πολιτικών ομάδων. Εγώ προσπαθώ να ε, σας δίνω το λόγο όσο το δυνατόν περισσότερο και με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία και να καταλήγω σε αποφάσεις αποδεκτές από όλους. Σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις. Νομίζω ότι θα ήταν δίκαιο όλοι να βοηθούμε να επιλύονται καταστάσεις όταν προκύπτουν να προσπαθούμε λοιπόν να διευκολύνουμε το χειρισμό καταστάσεων και να μην επιμένουμε σε τυπικά διαδικαστικά ζητήματα. Και αυτό το λέω και για να μην είναι η διαδικασία τόσο χρονοβόρα, αλλά και για να μην δυσκολεύεται και η Επιτροπή στο σύνολό της εργασίας της. Αλλά προτείνω να μας πει η νομική υπηρεσία για το νομικό υπόβαθρο τη απόφαση που έχουμε λάβει για το ζήτημα της τροπολογίας 17 με τη δυνατότητα ε, απόσυρσης τροπολογίας ε, που είχε ε, προταθεί, που είχε υποβληθεί. Από ό,τι κατάλαβα, παρατηρώντας τη ψηφοφορία, υπήρξε μία παρανόηση όχι μόνο από μία πολιτική ομάδα, αλλά από περισσότερες και από ό,τι κατάλαβα έλαβε τη σωστή απόφαση ο πρόεδρος υποβάλλοντας ε, στο εκλογικό σώμα μία ακόμη ψηφοφορία για να καταλάβουμε ακριβώς ε, ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Για μένα υπήρχε σαφέστατη παρανόηση. Yes, If that is the Αν αυτή είναι η σωστή ερμηνεία, Εντάξει, θα πρέπει να επαναλάβουμε την ψηφοφορία, αλλά όχι να αποσύρθει η τροπολογία, γιατί από ό,τι κατάλαβα, αυτή τη στιγμή έχουμε ψηφίσει μία ε, τροπολογία, δεν ανήκει σε κανέναν, ούτε σοσιαλδημοκράτη, ούτε σε κανέναν, ανήκει στην Επιτροπή. Υπήρξε λοιπόν ένα σφάλμα και θα έπρεπε γι' αυτό να ξαναψηφίσει η, Ευρωπα... Ε, να ξαναψηφίσει η Επιτροπή μα. Ε, ε, ε, έτσι τουλάχιστον το καταλαβαίνω και το ερμηνεύω εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθο μπορώ να πω και εγώ κάτι. Να σας πω πώς το καταλαβαίνω εγώ. Εσείς είπατε ότι έπρεπε να ξαναγίνει η ψηφοφορία γιατί υπήρξε παρανόηση στην πρώτη ψηφοφορία, που σημαίνει ότι είναι σαν να μην έγινε ποτέ η πρώτη ψηφοφορία και δίνει τη δυνατότητα έτσι σε μία ε, ε ομάδα να αποσύρει μία τροπολογία πριν γίνει δεύτερη ψηφοφορία. Τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ε, βοήθησε στη σαφήνεια της ε, ε, κατάστασης. Όχι, δεν βοήθησε, αλλά αυτό συνέβη. Uh, Περνάμε τώρα στα σχέδια γνωμοδότησης για την ε, απαλλαγή για το 2009, τμήμα 3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Μπουζούτιλ είναι ο εισηγητής. Υπάρχει μία τροπολογία Ψηφίζουμε την τροπολογία και μετά ψηφίζουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε λοιπόν στην, την τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικός. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται με 37 ψήφου υπέρ και μία ψήφο κατά. Και καμία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν η έκθεση. Περνάμε στην ε, επόμενη απαλλαγή για την εκτέλεση του προπολογισμού για το οικονομικό έτος 2009 και την υπηρεσία θεμελιωδών δικαιωμάτων. Υπάρχει μία τροπολογία. Α, δεν υπάρχουν τροπολογίες. Ωραία. Από ψηφίζουμε το κείμενο έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 37 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά. Εγκρίνεται και πάλι. Περνάμε τώρα στην τρίτη, στο τρίτο σχέδιο γνωμοδότησης για την απαλλαγή σε σχέση με το Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία για το Οικονομικό έτος 2009. Μία τροπολογία έχει υποβληθεί. Ψηφίζουμε την τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το, το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. σχέδιο γνωμοδότησης ε, για την εφαρμογή του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2009 και πάλι. Μία τροπολογία υπάρχει. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το τελικό κείμενο. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 37 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αστυνομικών, ε, πάλι του κυρίου Μπουσούτιλ. Έχουμε εδώ ε, κάποιες περισσότερες τροπολογίες. Ψηφίζουμε την πρώτη τροπολογία, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ όχι καταπίπτει η 9 η 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έναρξη. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομοφόνος. Ψηφίζουμε τώρα την απαλλαγή για το Frontex. Δύο τροπολογίες έχουν κατατεθεί. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ψηφίζουμε τώρα το κείμενο όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικός έναρξη ψηφοφορίας πέρας της ψηφοφορίας 37 υπέρ μία ψήφος κατά εγκρίνεται Περνάμε τώρα στο σχέδιο γνωμοδότησης ε, για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του άρθρου 10 των πρωτοκόλων ε, ε, πυροβόλων όπλων του ΟΗΕ για την αδειοδότηση εξαγωγών, εισαγωγών και προσωρινών μέτρων. Η κυρία Βερονίκ Ματιό είναι η συγγήτρια. Έχουμε κάποιες ε, τροπολογίες, ίσως η κυρία Ματιού να ήθελε να πει ορισμένα πράγματα πριν από την ψηφοφορία. Όχι. Ωραία, τότε περνάμε αμέσως στην ψηφοφορία. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Καλύτερα να ελέγξουμε ηλεκτρονικώς. Την τροπολογία 2. Έναρξη της ψηφοφορίας. Now the vote is closed. Πέρας. 20 against. 20 ε, κατά 17 ε, υπέρ. Άρα απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 22 κατά, 15 υπέρ, άρα απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο? Κυρία Αλβάρο, θέλετε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικός? Ωραία. Την 31 λοιπόν ψηφίζουμε ηλεκτρονικός, έναρξη ψηφοφορίας. Όχι, 31 είναι, λέει ο πρόεδρος. Α, είναι η 8 διορθώνει ο πρόεδρος, συγγνώμη. Την 8 λοιπόν ελέγχουμε ηλεκτρονικώς. Όχι, την 31 ή την 8. Μα ζητήσατε να ελεγχθεί η 31. Ωραία. Την 31 τότε. 25 κατά 13 υπέρ. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 8 τώρα. Υπέρ. κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 32. Θέλετε να ψηφίσουμε και πάλι την 8 ηλεκτρονικός. Εντάξει. Ηλεκτρονικός έλεγχος της 8. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 19 κατά 18 υπέρ. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Έχουμε δύο τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ.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 Θέλετε να την αποσύρετε? 38 τότε, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 39, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 19, υπέρ. Αποσύρεται. 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Η 20 αποσύρεται. 41 τότε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43. Α, συγγνώμη, 44 διορθώνει και 45 είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε ηλεκτρονικό τότε τη 44 και 45. Έναρξη ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 18 κατά, εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24, δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε, είναι γλωσσική ε, φύσεως. 25, υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται 26, υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. Η 47, υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται 27, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε τώρα το τελικό κείμενο ηλεκτρονικός έναρξη ψηφοφορίας πέρας 22 υπέρ, 14 κατά και 2 αποχές, οπότε εγκρίνεται. Ευχαριστούμε πολύ για την ψηφοφορία. Νομίζω τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Οπότε να περάσουμε στα επόμενα σημεία της ημερήσιας διάταξης.

point number 12 concerning the minimum Σημείο 12 σχετικό με τα ελάχιστα πρότυπα τι ελάχιστε απαιτήσει για τι διαδικασίε με τι οποίε τα κράτη-μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώ του πρόσφυγα. Αναδιατύπωση. Έχουμε μία έκθεση τη συναδέλφου κυρία Γιγιόμ και ε, θα πρέπει να ε, συζητήσουμε σχετικά με τις τροπολογίες. Είναι η τελική συζήτηση για τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν για την ε, διαδικασία περιδικασιών πριν από την συνεδρίασή μας που είχε προγραμματιστεί για τις 17 Μαρτίου. Η κυρία Γιγιόμ έκανε διάφορες διμερείς επαφές με τους σκιώδεις εισηγητές για να ε, διευκρινιστεί η διατύπωση των τροπολογιών και για να συζητηθούν οι συμβαστικέ προτάσεις. Θα ακούσουμε λοιπόν την εισηγήτριά μας, την κυρία Σιλβί Κιγιόμ, ώστε να μας αναφέρει ποια είναι τα αποτελέσματα των συζητήσεων με τους σκιώδεις εισηγητές και στη συνέχεια θα ακούσουμε τα μέλη καθώς επίσης και τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, την κυρία Μαριάλ ε, Καν. Η κυρία Γκυγιόμ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς δύο λόγια εισαγωγικά για να σας πω ότι το Κοινοβούλιο μπήκε στις συζητήσεις για τα διάφορα ε, νομοθετικά κείμενα που θα πρέπει να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή, Επιτροπή, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση για το άσυλο και ανάμεσα σε αυτόν τον μηχανισμό που είναι αρκετά πολύπλοκος, ε, έχουμε μια πρόσθετη απόφαση του δικαστηρίου που δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό και επιβεβαιώνει την θέση που είχαμε. Είναι μια απόφαση της 21ης Ιανουαρίου που ξέρετε ίσως και που επιβεβαιώνει πολλές θέσεις που σχετίζονται με τις προσωπικές ε, ε, συνεντεύξεις, με την ε, ανασταλτική ισχύ της αίτηση κλπ. Η απόφαση αυτή λοιπόν μας επιτρέπει να ξεκινήσουμε μια συζήτηση σχετικά με την ευαλωτότητα των ετούντων άσυλο. Είναι μια απόφαση αρκετά ε, σημαντική και διαφωτιστική και το κείμενο αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας για τους μελλοντικού μας ε, προσανατολισμούς. Για να έρθουμε τώρα πιο συγκεκριμένα στις πολυάριθμες πραγματικά τροπολογίες που υπέβαλαν οι συνάδελφοι, που εξέτασα με μεγάλη προσοχή, πρέπει να σας πω, ε, αλλά Πρέπει να σας πω επίσης, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι αρκετά πολύπλοκη υπόθεση να βρεθούν συμβαστικέ λύσεις, αν και κανείς ποτέ δεν θα πρέπει να απελπίζεται στη ζωή. Θα ήθελα να επιμείνω στην ανάγκη να διατηρηθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα και στην δικαιοσύνη, το, την ακρίβεια των διαδικασιών. Αυτό είναι το αντικείμενο των εργασιών μας. Και αυτή ακριβώς είναι η ισορροπία προς την οποία τίνει και το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επ' αυτού νομίζω ότι θα πρέπει ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε ώστε το κείμενο της Κομισιόν να λέει πράγματι αυτό που θέλει να πει και να μην το κάνουμε να λέει αυτά που δεν θέλει να πει. Για να αναφερθώ σε ορισμένες μόνο τροπολογίες, για να μην εξελίσω τώρα το θέμα, θέλω να σας πω ότι η πρόταση επιτρέπει την εξέταση της με την επιτυχημένη διαδικασία για συγκεκριμένε κατηγορίες ετούντων, το οποίο θα το συζητήσουμε αργότερα, αλλά πρέπει επίσης να πούμε ότι στη σημερινή δικασία προβλέπονται 22 λόγοι επιτάχυσης της διαδικασίας εξέτασης μια αίτησης. Πράγμα το οποίο πάει εντελώς αντίθετα προς την επιθυμία μας για εναρμόνιση και που ε, επίσης δημιουργεί αυτή, ε, αυτός ο μεγάλος αριθμός ε, ε, ε, ε αιτιολογήσεων διαφορετικές, οδηγεί σε διαφορετικές πρακτικές στα κράτη-μέλη. Κάτι άλλο που δεν λέει αυτή τη στιγμή το κείμενο της Κομισιόν και που έδωσε λαβή σε τροπολογίες είναι ότι αντίθετα από διάφορες εκτιμήσεις το κείμενο της Κομισιόν προβλέπει επίσης και μια υποχρέωση συνεργασίας του ετούντος την διεθνή προστασία συνεργασίας του δηλαδή με τις αρχές. Αντίθετα επίσης και με κάποιες άλλες εκτιμήσεις που επίσης οδήγησαν σε τροπολογίες, το κείμενο επιτρέπει να αποκαλύπτονται καταχρηστικές αιτήσει. Και αυτό γίνεται δυνατό χάρη σε αυξημένη ενημέρωση των ε, ανθρώπων που είναι αρμόδιοι για την εξέταση των ε, ε, αιτήσεων και που θα πρέπει να επιδεικνύουν τις αποδείξεις. Επίσης, για άτομα που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, αντίθετα από ό,τι διάβασα, δεν προβλέπεται για τους ιδιαίτερα ε, καταπονημένους ε, τούντες, ε, που έχουν υποστεί βασανιστήρια και που μερικές φορές δεν είναι, δεν είναι σε θέση να εκφραστούν για να ζητήσουν προστασία. Και αυτό ενισχύει την ανάγκη των συναντήσεων και των συναντεύξεων. Όλα αυτά πιστεύω ότι δημιουργούν μια λογική που δεν μας παραπέμπει σε απλή πρόσθεση των επιμέρους εθνικών πρακτικών. Το σημερινό μου σύστημα διατηρεί πολλές διαφορές όσον αφορά την επιτυχημένη διαδικασία και άλλα ε, που είναι ένα σύστημα ασύμβατο με ένα ενιαίο καθεστώς που θα πρέπει να ισχύει σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποτελεί τις κατευθυντήριες γραμμές για το καθένα από τα κράτη-μέλη. Κλείνω κύριε Πρόεδρε γιατί δεν μπορώ να αναφερθώ σε στο σύνολο όλων των τροπολογιών που υποβλήθηκαν. Θα ήθελα λοιπόν να τελειώσω αναφερόμενοι σε τέσσερα σημεία που μου φαίνονται σημαντικά και που θα συζητήσω με τους σκιώδες. Το ένα σημείο το οποίο μου φαίνεται σημαντικό είναι το δικαίωμα για προσωπική συνέντευξη. Είναι πραγματικά μια προτεραιότητα που θα πρέπει να υπερασπιστούμε. Και αν ε, υπάρχουν εξαιρέσεις, ε, θα πρέπει να υπάρχουν μόνο σε πολύ στενά καθορισμένα πλαίσια, όπως προβλέπεται και από την ε, υφιστάμενη πρόταση. Δεύτερον, θα πρέπει να υποστηρίξουμε την Κομισιόν την πρότασή της σχετικά με τις ε, αρμοδιότητες των ε, υπηρεσιών, των αρχών. Ε, τρίτον, θα πρέπει ένας ετών να είναι σε θέση να αμφισβητήσει την έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας και θα πρέπει γενικά να δούμε αυτή την έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας και της ασφαλούς χώρας προέλευσης και θα πρέπει να πιέσουμε για να αποκτήσουμε ένα ευρωπαϊκό κατάλογο ασφαλών ε, χωρών. Ε, από την άλλη μεριά, πράγμα το οποίο μου φαίνεται εντελώς ε, αντιφατικό. Κάτι άλλο, η δυνατότητα εκπροσώπησης είναι μια επιπλέον εγγύηση που θα πρέπει να ε, προωθήσουμε λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος ε, των αιτήσεων ασύλου, κάτι το οποίο βλέπω κάθε μέρα στη δουλειά μου θα πρέπει να επιμείνουμε εδώ, πιστεύω, γιατί αυτό είναι ε, προ το όφελο του ετούντο αλλά και του κράτου, το οποίο θα μπορούσε πολύ εύκολα και γρήγορα να εντοπίσει τι ανάγκε προστασία, αλλά και επίση να απορρίπτει τι αιτήσει που είναι καθαρά καταχρηστικέ. Και αυτό επίση θα οδηγήσει ε, στο front loading ε, της Κομισιόν. Αυτά πολύ γρήγορα κύριε Πρόεδρε ήθελα να πω για την κατάσταση στην οποία έχει φτάσει η συζήτηση για το θέμα αυτό με όλες τις σχετικές δυσκολίες. Οι εργασίες όμως συνεχίζονται. Ευχαριστώ κυρία Γκυγιόμ. Ίσως θα μπορούσαμε να δώσουμε το λόγο στην ε, Κομισιόν, στην κυρία Μυριέλ Κον, πριν να αρχίσουμε την ε, γενική συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής μας. Η εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω την Σιλβί Γκυγιόμ για την ε, σύνοψη αυτή που έκανε και που πραγματικά ανταποκρίνεται στην φιλοσοφία της πρότασης της Κομισιόν. Εμείς βλέπουμε βεβαίω ότι όλες αυτές οι, τροπολα... οι τροπολογίες αποδεικνύουν τη δέσμευση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκ μέρους όλων των ομάδων, ε, σε σχέση με την οδηγία αυτή που έχει σε σκοπό να έρθουμε σε μια δεύτερη φάση της εναρμόνισης πριν από το τέλος του 2012 ε, σε μια οδηγία που θα, είναι, θα έχει πραγματικά προστιθέμενη αξία σε σχέση με το σημερινό και εκτιμένο. Και ιδιαίτερα ε, στην διευκρίνηση ορισμένων ενιών και στην ποιότητα των διαδικασιών σε πρώτο επίπεδο ε, την επένδυση σε αυτή την πρώτη περίοδο που είναι κρίσιμη για τους ε, ετούντες ε, άσυλο. Είναι κάτι το οποίο θα δώσει και αποδίδει ήδη στα κράτη-μέλη που επενδύουν σε αυτό το πρώτο μέρος της διαδικασίας και έχουμε τις αποδείξεις. Όπως ξέρετε η Κομισιόν έχει δεσμευτεί να υποβάλει μια πρόταση αναθεωρημένη σε σχέση με την περσινή της, γιατί γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια δύσκολη συζήτηση και θέλουμε να συμβάλλουμε στην επίτευξη ε, κοινών στόχων μεταξύ όλων των ε, συνομοθετών πριν από το τέλος του 2012. Για το λόγο αυτό ακριβώς οι θέσεις του Κοινοβουλίου είναι ε, ένας παράγοντας κλειδί για μας ε, θα έχουμε και άλλες συναντήσεις με την εισηγήτρια μέχρι την επόμενη συνεδρίασή σας για να διευκρινίσουμε μερικά ακόμα σημεία της πρότασης αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην ε, κάνουμε ε, την πρόταση της Κομισιόν να λέει πράγματα που δεν θέλει να πει. Εν πάση περιπτώσει, όπως το ανέφερε η κυρία Γιγιόμ, ένα σημείο αναφοράς για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την αναθεωρημένη της πρόταση θα είναι οι μεγάλες τάσεις της ευρωπαϊκής νομολογίας. Είτε πρόκειται για το δικαστήριο του Στρασβούργου είτε για αυτό του Λουξεμβούργου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκάν. Να δώσω τώρα το λόγο του στα μέλη της ε, Επιτροπής. Στη συζήτηση. Κυρία Βέμπερ, θέλετε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Επόσον όλοι μιλάνε γαλλικά, αισθάνομαι ότι και εγώ πρέπει να τα πω γαλλικά. Εγώ θα ήθελα να πω για το θέμα αυτό, δεν είμαι βέβαια σκέωδης εισηγήτρια, αλλά θα ήθελα να πω ότι η ομάδα των φιλελευθέρων και δημοκρατών ε, είναι ε, ιδιαίτερως ικανοποιημένη γιατί θα προχωρήσουμε επιτέλους ε, με τις ε, διαδικασίες για το ζήτημα αυτό. Γνωρίζουμε ότι έχουν υποβληθεί πολλές τροπολογίες και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μία γραμμή ε, της ομάδος σε σχέση με τις τροπολογίες που θέλουμε πραγματικά να υποστηρίξουμε και τις τροπολογίες που κατά πάσα πιθανότητα θα απορρίψουμε αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό κατά τις δύο ερχόμενες εβδομάδες πριν την ψηφοφορία δηλαδή θα είναι να καταφέρουμε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και στη συνέχεια ευρύτερα στο Κοινοβούλιο όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνένεση. Γιατί κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποσταλεί ένα μήνυμα στο Συμβούλιο, ένα πολύ ισχυρό μήνυμα από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που, ότι θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε και να προχωρήσουμε με τα μέτρα που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν κάποιες ιδέες, κάποιες τροπολογίες που θέλουμε πραγματικά να υποστηρίξουμε, αλλά νομίζω ότι για την ώρα θα αρκεστώ στο να πω ότι κατά τις ερχόμενες δύο εβδομάδες πρέπει να διαπραγματευτούμε πάρα πολύ μεταξύ μας για να καταφέρουμε να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερη η υποστήριξη του ζητήματος αυτού και στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο ευρύτερα. Γιατί αν δεν καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό, νομίζω ότι το Συμβούλιο θα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένο γιατί θα βρίσκεται σε μια πραγματικά ισχυρή ε, θέση κατά της συγκεκριμένης πρότασης. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χολμάιερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς είναι πολύ σωστή η παρασύρηση ότι θα πρέπει να έχει το δικαίωμα σε προσωπική συνομιλία κάθε ένας που αιτείται το άσυλο, βεβαίως με διερμηνέα Ως προσθέτω, το θέμα της ε, προσφοράς νομικής ε, βοήθειας είναι η εξέλιξη της συζήτησης όπως ε, τη βλέπω τώρα τέτοια που μας οδηγεί σε επιβάρυνση οικονομική υπερβολική για τα κράτη. Και ως εκ τούτου δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει δυνατότητα για πλήρη νομική υποστήριξη σε κάθε περίπτωση. Μπορούμε να τα συστήσουμε όμως αυτά. Μην ξεχνάμε ότι αν φτάσουν σε ένα κράτος ε, μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα 100.000 ετούντας στο άσυλο, θα είναι μάλλον αδύνατο για το κράτος αυτό να καλύψει, τουλάχιστον για τα περισσότερα, να καλύψει αυτά τα έξοδα. Λαμβάνοντα υπόψη λοιπόν αυτή την προοπτική, αυτή, την πιθανότητα, παρακαλώ του συναδέλφου να δείξουν κατανόηση. Επίσης για την ε, ε, ταχεία απονομή ή ταχεία διαδικασία. Θα ήθελα να πω το εξή. Η Επιτροπή φαίνεται ότι απορρίπτει την ιδέα αυτή εάν δεν αποτελεί κίνδυνο, εάν αποτελεί κίνδυνο μάλλον για την ασφάλεια ο ετών το άσυλο, για την εθνική ασφάλεια κτλ. εγώ θεωρώ ότι έχει νόημα σε τέτοια περίπτωση κινδύνου δηλαδή για την εθνική ασφάλεια η ταχεία διαδικασία. Επίσης, θα ήταν καλό πιστεύω να σκεφτούμε σε περίπτωση όπου κάποιος έχει υποβάλει αίτηση ασύλου με ε, δεδομένα ή δηλώσεις ε, τελείως ασυνάρτητες, αβάσιμε, προφανώς αβάσιμες κτλ. Γιατί να μην υπάρχει ζήτημα ταχεία διαδικασίας. Μην ξεχνάμε ότι σημαντικό μερίδιο εκείνων το, οι οποίοι ζητούν το άσυλο ε, προβαίνουν σε αυτή την κίνηση για άλλους λόγους και όχι γιατί, γιατί χρειάζονται τέτοια προστασία ασύλου. Επίσης, στις ακόλουθες αιτήσει λεγόμενα, επακόλουθες αιτήσει. Όταν ε, εξαφανίζεται κανεί, ε, βγαίνει στην παρανομία κτλ., θα πρέπει να σταματάει αυτή η διαδικασία. Έτσι ώστε να μπορεί να επαναληφθεί ή να επανεκκινηθεί σε περίπτωση που αυτό ξαναεμφανιστεί. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν ε, το έχω βρει εγώ, μια πρόταση που έχω βρει εγώ, αλλά που έχω ακούσει από νομικού. Και γι' αυτό νομίζω θα ήταν καλό σε τι περιπτώσει επακόλουθων αιτήσεων να υπάρχει η δυνατότητα για πλήρη εξέταση αυτής της ετάσης ε, της μια διαδικασία έστω όχι ε, ταχεία, έστω και αν δεν υπάρχουν νέοι λόγοι που προβάλλονται. Και επίσης, ενδιαφέρον νομίζω το να δούμε τι είδους ε, συνέπειες μπορεί να έχει ένα κράτος μέλος το οποίο δεν εφαρμόζει πλήρως την νομοθεσία αυτή. Το έχουμε ξαναδεί φυσικά, αλλά ιδιαίτερα στο θέμα του ασύλου έχει μεγάλη σημασία και το Κοινοβούλιο έχει νομίζω κάθε λόγο να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή από τα 27 κράτη-μέλη του δικαίου του σχετικού με το άσυλο. Αυτά και κατά τα άλλα πιο πολύ ε, ευχές βλέπουν να το μέσα στο κείμενο παρά διατάξεις. Thank Ευχαριστώ πολύ κυρία Χολμάιερ. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο? Δεν θέλει κανείς ε, να σχολιάσει την παρουσίαση της ε, εισηγήτριας, κυρίας Γιγιόμ. Οπότε, κυρία Γιγιόμ, σας ξαναδίνω το λόγο, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Πάρα πολύ σύντομα, γιατί ανέφερα προηγουμένως αυτό που ήταν ε, πάρα πολύ σημαντικό για τις ε, συζητήσεις μας ε, και στο πλαίσιο της είπα της αρμοστίας του ΟΗΕ η κυρία Χολμάιρ γνωρίζει ήδη τα τρία τέταρτα του ζητήματος και το ένα τέταρτο θα το συζητήσουμε κατά τις επόμενες εβδομάδες δύο, δύο ακόμη ζητήματα μου φαίνονται σημαντικά για τις συζητήσεις μας είναι λίγο περίεργη η χρονική στιγμή γιατί υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή λόγω των ανατροπών γύρω από την λεκάνη της Μεσογείου και είναι γεγονός ε, ότι υπάρχουν ε, διάφορες ε, προτάσεις ε, στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής, ανάκλησης διεθνούς προστασίας και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί λένε ότι είναι πιο σημαντική η κίνηση από, από Ανατολή προς Δύση από ότι από τον Νότο προς το Βορρά. Αλλά αυτή η υπόθεση έκρηξης της ε, των μεταναστευτικών ροών ε, δεν μπορεί να την εκμεταλλευτούμε ε, λόγω της πίεσης για να καταλήξουν επιτέλους σε κάποια συμφωνία τόσο σημαντικά ζητήματα νομίζω ότι είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τη δυνατότητα να αιτείται ε, κάποιος ε, άσυλο παρά τη δύσκολη κατάσταση και τις πιέσεις. Σε σχέση με το θέμα που αναφέρατε προηγουμένως, ε, και το, κατά το πώς, αν υπάρξει αναθεωρημένη πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς θα τοποθετηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, εγώ για να απαντήσω στο ερώτημα αυτό, θα έλεγα το εξής είναι ότι η τοποθέτηση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί από αυτούς ε, τους ε, προσανατολισμούς ε, θα έχουμε και τη νέα διάρθρωση του κειμένου. Εγώ θα ήθελα όμως να έχουμε ένα φιλόδοξο κείμενο το οποίο θα μπορέσουμε να υπερασπιστούμε. Δεν μιλάμε μόνο για σύμβολα. Εγώ ελπίζω ότι είναι ακριβώς αυτό που συνιστά το ρόλο μας του συνομοθέτη και είναι μια, μια δυνατότητα να το... να το αποδείξουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτός είναι πολύ σημαντικός, ε, γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος μας στη συζήτηση αυτή. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε το σημείο 13 σε σχέση με την εντολή για τον τριμερή διάλογο για το ε, σχέδιο προπολογισμού του 2012. Θα κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Έχουμε εδώ τη συναρφό Φραντσέσκα Βαλτσάνη, υπεύθυνη για τον προπολογισμό. Και έτσι μπορούμε να κάνουμε την πρώτη συζήτηση για τον προπολογισμό 2012 στην Επιτροπή μας. Κυρία Βαλτσάνη, λοιπόν, αρμόδια για τον προπολογισμό. συναντάται με τις ε, ειδικές κοινοβουλευτικές επιτροπές για να συζητήσει σε κάθε περίπτωση τα θέματα του προπολογισμού τους. Η Επιτροπή μας δεν έχει ορίσει ε, συντάκτη γνωμοδότηση για τον προπολογισμό. Η έκθεση θα δημοσιευθεί τον Απρίλιο, στις 20 Απριλίου και συζήτησαν ε, στόχο έχει να εξασφαλίσει μια ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα αυτά. Ας ακούσουμε τώρα την κυρία Παλτσάνη. Και μετά τους άλλους βουλευτές που ενδεχομένως θέλουν να λάβουν το λόγο. Κυρία Παλτσάνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή είναι μια πρώτη συνάντηση με, τις πρώτες, με την πρώτη από τις ε, ειδικέ ε, επιτροπές και είναι μια φάση που τη θεωρώ πολύ σημαντική για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων για τον προπολογισμό του 2012. Φέτος πραγματικά η πρότασή μου είναι κάτι το καινούριο. Θέλουμε να αξιολογήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό μια μεγάλη καινοτομία που για πρώτη φορά ε, κάνει ε, ένα πραγματικά ε, βήμα προς τα μπροστά για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Για πρώτη φορά ε, φέτος τα εθνικά κοινοβούλια θα προσπαθήσουν να καταστήσουν συνεπεί στους προϋπολογισμούς τους με, την, με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. πρόκειται για το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Αυτό μα οδηγεί στη θετική του 2020 που θέλει να είμαστε συνεπείς και να έχουμε κοινού στόχου. Και αυτή η πρώτη ευκαιρία πρέπει να αξιοποιηθεί πιστεύω γιατί μας επιτρέπει να επιτύχουμε πολλούς στόχους. Μας επιτρέπει να είμαστε πιο, ε, πιο αξιόπιστοι, πιο ισχυροί, να αξιοποιήσουμε περισσότερο τους διαθέσιμους πόρου σε μια στιγμή κρίση και ε, μας επιτρέπει να... Ε, προσφέρουμε αυτή την προστιθέμενη αξία σε αυτό το πολύ σημαντικό άξονα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, ε, το κρίσιμο σημείο για να έχουμε έναν προϋπολογισμό συνεπή με τη στρατηγική του 2020 και με το ευρωπαϊκό εξάμεινο που θέλει πραγματικά να επιτύχει τη συνοχή ανάμεσα στους εθνικούς και τους ευρωπαϊκούς στόχους πρέπει να είναι ακριβώς το μεγάλο πλαίσιο ε, για την επόμενη χρονική περίοδο που θα πρέπει να έχει πέντε στόχους. Όχι μόνο αυτούς που πρότεινε η Κομισιόν, αλλά και αυτούς που το Κοινοβούλιο με τα ψηφίσματά του έχει υιοθετήσει ε, θερμά. Η στρατηγική του 2020 είναι ιδιαίτερα σημαντική για αυτή την Επιτροπή πάνω απ' όλα γιατί ένας από τους στόχους, η καταπολέμηση δηλαδή της φτώχειας και η μεγαλύτερη ε, κοινωνική ενσωμάτωση, είναι πραγματικά ο κύριος άξονας όλων των προγραμμάτων ε, και των πρωτοβουλειών που ανήκουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Όπως ε, πρόκειται και για μια ευληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής, η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα δηλαδή κατά της φτώχειας. Άρα πιστεύω ότι το να προσπαθήσουμε να, επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας για τον προβλησμό του 2012, ούτως ώστε να αναδειχθεί σαφώς αυτή η ιδέα που έχουμε όλοι, ξεκινώντας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο μέχρι όλα τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δηλαδή, η βούλησή μας να έχουμε μια πραγματική στρατηγική που θα αποφεύγει τα λάθη του, παρελθό, του παρελθόντος και αν θέλουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτούς τους μεγάλους κοινού στόχους που είναι προτεραιότητα όχι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή εδώ έχει η ειδική αρμοδιότητα για τον τομέα 3α του προϋπολογισμού που από το 2007 αυξήθηκαν οι διαθέσιμοι πόροι για, αυτή, για αυτόν τον τομέα. Αλλά υπάρχουν και πολλοί οργανισμοί που εμπίπτουν σε αυτόν τον τομέα. Οκτώ ε, και που απορροφούν περίπου το 22% όλων των διαθέσιμων κονδυλίων αυτού του τομέα. Ένας τομέας που σίγουρα περιλαμβάνει στόχους που είναι, έχουν μεγάλη σημασία για τη στρατηγική του 2020 και θα αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις. Και αναφέρομαι ιδίως στα πρόσφατα γεγονότα της Τινησίας, της Αιγύπτου και της Λιβύης. Πρόκειται για ένα τομέα του προϋπολογισμού που θα πρέπει να ανταποκριθεί σε απαιτήσει που δύσκολα θα μπορούσαμε να φανταστούμε στο παρελθόν. Το περιθώριο που σήμερα προβλέπεται από το δημοσιομικό έγγραφο, που είναι το πρώτο βήμα για αυτή τη διαδικασία του προϋπολογισμού, είναι ε, μειωμένο σε σχέση με το ε, περιθώριο που υπήρχε σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2011. Ε, Έχουμε 26 εκατομμύρια σε σχέση με τα 77. Είναι όμως μεγαλύτερο περιθώριο από αυτό που προβλεπόταν στο προγραμματισμό της περσινής χρονιάς. Πρόκειται ένα περιθώριο ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί ε, από αυτό εξαρτάται ε, τι περιθώρια υπάρχουν για ε, πιλωτικά προγράμματα, για πρωτοβουλίες και πολιτικές στα πλαίσια αυτού του τομέα του προϋπολογισμού. Αυτό το περιθώριο λοιπόν, που είναι ε, εν τέλει ίσως ε, ανεπαρκές για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, στα πλαίσια λοιπόν αυτού του περιθωρίου θα πρέπει να επαναπροτείνουμε δύο από τα ε, αιτήματα που ε, έχετε δει ήδη στο έγγραφο εργασίας. Το πρώτο αφορά την ανάγκη να γίνει πιο συνεκτική η προσπάθειά μας με, στα πλαίσια της ε, στρατηγικής του 2020 και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και πρόκειται για, για τον καθορισμό των τομέων που έχουν προτεραιότητα σε σχέση με την υλοποίηση της στρατηγικής του 2020. Αλλά παράλληλα υπάρχει και το αντίθετο αίτημα. Αν θέλουμε να δώσουμε μια πραγματική ευελιξία στον προϋπολογισμό και να τον κάνουμε ένα εργαλείο που θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις πάντα νέες μας στις όλο και, ε, πιο, ε, και σε όλο και διαφορετικές προτεραιότητές μας, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επαναπροσδιορισμού των ε, προτεραιοτήτων. Ε, να δούμε αν υπάρχουν αρνητικές προτεραιότητες. Γιατί και αυτό η αναθεώρηση των προτεραιοτήτων είναι ένας τρόπος ανάληψης νέων δράσεων. Για να τα κάνουμε όλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε ήδη από τώρα να και να προσδιορίσουμε ποιε δράσεις έχουν στρατηγική σημασία και ίσως θα πρέπει να ενισχυθούν και να αυξηθούν το 2012 και ποιε καινοτομίε και αναφέρομαι στα πιλωτικά ε, προγράμματα και προπαρασκευαστικέ δράσει θα πρέπει να ενισχυθούν ή να διατηρηθούν. Επίση, θα πρέπει να κάνουμε μία ανάλυση σχετικά με το πώ λειτουργήσαν ε, ε, τα πιλωτικά προγράμματα και οι προπαρασκευαστικέ δράσει που λειτουργούν ήδη. Γιατί μας επιτρέπει κάτι τέτοιο να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα του μέσου που έχει επιλεγεί και άρα να προβλέψουμε μια αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και για το μέλλον. Στην Επιτροπή εδώ υπάρχει ένα έγγραφο εργασίας που έχει την πρόθεση να λειτουργήσει σαν αφορμή για να ξεκινήσει μια συζήτηση ε, για όλους αυτούς τους στόχους που δεν είναι, παραλαμβάνω, στόχοι του Κοινοβουλίου που ε, καθορίζονται ε, χρόνο με το χρόνο. Πρόκειται για τους στόχους του ευρύτερου πλαισίου της Ευρώπης του 2020. Και το έγγραφο αυτό πέραν μάλλον του εγγράφου αυτού, έχω υποβάλει και μια πρόταση ε, ψηφίσματος. Διότι οι προτάσει του Συμβουλίου φέτος είναι ιδιαίτερα λεπτομέρειες και γι' αυτό πίστευσα, θεώρησα σκόπιμο να δώσουμε κι εμείς μια απάντηση. Στην πρόταση ψηφίσματος θα δείτε ότι προτείνω ε, επειδή υπάρχει αυτή η ανοιχτή συζήτηση ε, με τις διάφορες επιτροπές, να αφήσουμε ανοιχτό το θέμα του καθορισμού των ε, τομεακών προτεραιοτήτων, που είναι ένα λεπτό θέμα, να δούμε μόνο ποιες είναι οι μεγάλες προτεραιότητες που θέλει να θέσει το Κοινοβούλιο για το 2012 και σε σχέση και με τη στρατηγική του 2020 να τονίσουμε το θέμα της εργασίας που περιλαμβάνεται σαν στόχος και στην Ευρώπη του 2020, μια Ευρώπη δηλαδή με μεγαλύτερη απασχόληση, με περισσότερες επενδύσεις, όχι μόνο για την έρευνα και την ανάπτυξη, αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι ένα ε, θεμελιώδης βήμα λοιπόν αυτό στην Επιτροπή μας για τον προσδιορισμό των ειδικών προτεραιοτήτων που θα έπρεπε να χρησιμεύσουν για έναν επικοδομητικό διάλογο που θα έχουμε και με τα Εθνικά Κοινοβούλια από τις 13 Απριλίου και μετά. Ούτω ώστε το Κοινοβούλιο μας να ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής του 2020 που θέλουμε να γίνει μια πραγματικότητα χρήσιμη για τους ε, συμπολίτε μας κατά τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την Βαλτσάνη σε ακούσουμε τώρα και τους βουλευτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και την εισηγήτρια που βέβαια βρήκε χρόνο να έρθει σε εμά. Να μας κάνει αυτή τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίαση και να ακούσει τις παρατηρήσεις μας. Φαντάζομαι ότι κάθε μία από τις επιτροπές που επισκέπτεται τις λένε λέει ότι έχει πάρα πολύ σημαντικό για τα ζητήματα του προπολογισμού πεδίο αρμοδιοτήτων και θα την απογοητεύσω και εμεί το ίδιο πράγμα θα πούμε. Και εμεί πιστεύουμε ότι οι αρμοδιότητε τη Επιτροπή μα έχουν άκρα σημασία και αξίζουν άκρα προσοχής, για τον προπολογισμό του 2012. Και πέραν αυτού θα ήθελα να πω ότι οι επιλογές για τον προπολογισμό του 2012 θα πρέπει να δώσουν τον τόνο για τις προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές. Έχουν αυτή τη σημασία. Και περιμένω να κάνουμε σε Πεδολίμπε πολύ σύντομα συζήτηση για τις δημοσιονομικές προοπτικές και πώς μπορούμε να τις ε, εξετάσουμε υπό την έποψη της ελευθερίας, δικαιοσύνης και προστασία των πολιτών και νομίζω ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ιδιαίτερο το επόμενο βήμα για την Ένωση είναι ακριβώς να μετατραπεί σε ένωση των πολιτών. Οι πολίτες πρέπει να αποτελούν το σημείο εστίασης της ένωσης μας. Αυτό το πολιτικό μήνυμα πρέπει να αποσταλεί, να μεταφερθεί στους συναδέλφους μας από την Επιτροπή των Προπολογισμών. Πολλά είναι τα ιδιαίτερα θέματα που έχω υπόψη μου όσον αφορά τον προπολογισμό του 2012. Φερρυπίν, τα τέσσερα πρόγραμμα για τη μετανάστευση και την αλληλεγγύη δικής μας αρμοδιότητας. Δυστυχώ, ακόμη δεν έχει προχωρήσει η μέσω προθεσμή αναθεώρηση αυτών των προγραμμάτων, την οποία θα ήταν χρήσιμο να έχουμε. Το ταχύτερο δυνατό για να μπορέσουμε να σχολιάσουμε πιο συγκεκριμένα τι θέλουμε για τον προπολογισμό του 2012. Τέσσερα σημαντικά λοιπόν προγράμματα. Και ένα άλλο θέμα Τελευταίε εξέλιξει, πρόσφατες εξελίξεις που έθεξε ήδη η συγγήτρια, ήταν στην περιοχή της Μεσογείου και οι οποίες μπορούν να προξενήσουν κύμα μετανάστευσης που δεν έχει δει μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο του χρειάζεται να αναλάβουμε δράση. Και απαιτείται επίσης να προβλεφθούν και σχετικοί πόροι για να αναλάβουμε δράση. Γιατί καλές είναι οι πολιτικές δηλώσεις, αλλά χρειάζεται να είμαστε σε θέση και να διαθέσουμε τους απαραίτητους ε, πόρους, χρηματοοικονομικούς πόρους, ώστε αυτές τις δηλώσεις μας να τις στηρίζουμε και με συγκεκριμένε πράξεις. Έχουμε επίσης ε, υπό το πεδίο αρμοδιότητων της Επιτροπής μας και το θέμα των υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες που ανήκουν στι δικέ μα αρμοδιότητες και καλό θα ήταν, Πρόεδρε, να μα πούν οι τα ηθήνοντα στελέχη αυτών των υπηρεσιών, τι σκοπού έχουν το 2012, τι θέλουν να κάνουν έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένε προστάσει προ την Επιτροπή των Προπολογισμών. Πάντως η Frontex, που είναι η πρώτη ε, αποκεντρωμένη υπηρεσία που ε, σκέφτεται κανεί στην Λίμπε, και ξεκινάει μια μεγάλη κλίμακα επιχείρηση στη Μεσόγειο δεδομένων των εξελίξεων σε χώρες όπως η Τινησία και η Λιβύη. Μια άλλη υπηρεσία η υπηρεσία στήριξης του ασύλου ξεκινά, είναι έτοιμη να ξεκινήσει επιχειρήσεις, οι οποίες όμως ε, ακόμη δεν έχουν αρχίσει. Το 2011 θα αρχίσουν και άρα χρειάζεται και μια πρόβλεψη για την εφαρμογή του προπολογισμού του 2012 πιστεύουμε θα έχει αναπτύξει πλήρω δραστηριότητέ τη. Τέλει για τελικά προγράμματα και προπαρασκευαστικέ δράσει. Νομίζω πρώτα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα δώσει στοιχεία με μια έκθεση για τον τρόπο με τον οποίο δράσεις που ήδη έχουν συμπεριληφθεί στον προπολογισμό του 2011 ε, υλοποιούνται. Πώς δηλαδή τις παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να μπορούμε να ε, προγραμματίσουμε για το επόμενο έτος. Ευχαριστώ τον κύριο Βοσούτελ. Θέλει κάποιο άλλο να λάβει το λόγο. Άλλε παρατηρήσει. Κυρία Κέλλερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντω θα πρέπει να κοιτάξουμε τι γραμμέ εκείνε του προπολογισμού όπου έχουμε ζητήματα αρμοδιότητα τη ε, ΛΥΜΠΕ με τη νέα συνθήκη, εν πάση περιπτώσει τη ε, Λισαβόνα δεν είναι και τόσο καινούριες πια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επίση κάτι άλλο που επίση συνθήκη νωρίτερα πιστεύω. Πριν να προσδιοριστούν νέε προτεραιότητε, καλό θα είναι να δούμε τι μα έχουν προσφέρει παλαιότερε αρμοδιότητε πριν να ξεκινήσουμε νέα σχέδια. Καλό θα είναι να δούμε τι αντίκτυπο είχαν τα παλαιά. τι πήγε καλά, τι δεν πήγε, τι έφερε αποτελέσματα και τι Γι' αυτό λυπούμε που έρχονται πάντα με τόση καθυστέρηση αυτές οι μεσοπρόθεσμε εκθέσει. Και έρχονται τελικά και ατελεί δεν είναι πλήρη. Γι' αυτό θα ήθελα να δω και μια τελική φάση ενό σχεδίου. Όπω είπατε, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν θέλουμε να τα διατηρήσουμε ή τι θέλουμε να τα κάνουμε. Για τα πιλωτικά σχέδια δεν είναι πάντα σαφέ ε, τι μοίρα έχουν. Θα αποφασίζουμε, θα το προωθούμε σε εφαρμογή και τελικά δεν ξέρουμε τι αποτέλεσμα φέρνουν. Ενώ θα θέλαμε να έχουμε μια σαφή αξιολόγηση για να δούμε αν πράγματι φέρνουν τα αποτέλεσματα που θέλουν. Ή αν πρέπει να ανταλλαγούν, να αντικατασταθούν από κάποια άλλα. Και εν πάση περιπτώσει χρήματα πιο πολλά μάλλον δεν θα έχουμε για τον χρόνο, γι' αυτό καλό θα ήταν να προσδιορίσουμε προτεραιότητες και να αποφύγουμε τις περιπτώσεις που έχουμε μέχρι τώρα να δίνουμε λεφτά σε σχέδια που δεν φέρουν αποτελέσματα τελικά. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κάτι άλλο. Όχι. Κάποια τελικά σχόλια, παρακαλώ, κυρία Μπαλτσάνη. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Νομίζω ότι καταλαβαίνω τις πολλές δίκαιες ε, ε, ανησυχίες που υπάρχουν ότι θα έπρεπε οι νέες ε, προτεραιότητες να συμβαδίζουν με δράσεις για τις οποίες υπάρχει μια κάποια βεβαιότητα για την αποτελεσματικότητά τους. Ιδιαίτερα θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στα πιλωτικά προγράμματα, ε, στα πιλωτικά έργα και στις προπαρασκευαστικές δράσεις, γιατί έχουν μια πραγματικά μεγάλη δυνατότητα να ε, δοθεί ε, μια νέα όθηση στον προϋπολογισμό αυτό το πακέτο ε, δεσμεύεται με προθεσμίες ε, που είναι πολύ κοντινές. Θα πρέπει να κάνουμε πολύ σύντομα την αξιολόγησή μας και άρα θα πρέπει να αξιολογήσουμε ε, ό,τι λειτουργεί ήδη πριν προτείνουμε νέες τέτοιες δράσεις για να καταλάβουμε ακριβώς σε ποιο βαθμό έχουν αποδώσει και κατά πόσο μπορούμε να βασιστούμε και στο μέλλον πάνω σε αυτές τις δράσεις και τα πιλωτικά προγράμματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πατσάνη νομίζω ότι συμφωνούμε ότι αυτό θα είναι το τελικό σχόλιο για αυτό το θέμα. Και τώρα... Θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι πρέπει να ορίσουμε σύντομα τον ε, εισηγητή για την Επιτροπή μας, για τον προπολογισμό, αλλά θα πρέπει να ετοιμαστούμε και για τη γνωμοδότησή μας που θα πρέπει να υποβληθεί στον τριμερή, για τον τριμερή διάλογο τον Ιούνιο για τον προπολογισμό. Και πρέπει να εγκριθεί μάλλον μέχρι το τέλη Μαΐου. Αυτό ήταν για το 13. Προς το παρόν πάμε στο 14. Ασφάλεια των αερίων μεταφορών με ειδική έμφαση στους σαρωτές ασφαλείας. Γνωμοδότηση του συνάδελφου που είναι υπεύθυνο από την Επιτροπή των Μεταφορών, τον κύριο Λουίς Δεγράντες, σχέδιο γνωμοδότησης. Όπως είπα, πρόκειται για την έκθεση για την ε, ασφάλεια των αέριων μεταφορών ε, με τη συνήθεια διαδικασία γνωμοδότηση, αλλά ζητήσαμε εμείς ε, να συμμετάσχουμε με τη διαδικασία του άρθρου 54, αλλά δεν εγκρίθηκε αυτό. Του 50 μάλλον, ή 51. Θα ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Δεγράντε και μετά την κυρία Σαρτζεντίνη. Κυρία Ντεγράντες, αν θέλετε να ξεκινήσετε με την παρουσίαση τη νομοδότησή σα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω μια αντίρρηση. Αν και δεν είμαι αρμόδιος για τη γνωμοδότηση, απλώς εκ μέρους της ομάδας μου παρακολουθώ την έκθεση της κυρίας Σαρτζεντίνη. Επομένω, η σειρά μάλλον δεν είναι σωστή. Ίσως είναι σκοπιμό το να ξεκινήσει η κυρία Σαρτζεντίνη που έχει την αρμοδιότητα για την έκθεση. Και όταν έρθει η ώρα μου, μιλώ και εγώ εκ μόνος τη μου. Καλώ, κυρία Σαρτζεντίνη, Όσο συντάξει νομοθέτηση, έχετε το λόγο. Είχα ήδη κάπως μπερδευτεί. Όπως είπατε, η έκθεση αυτή δεν θα πρέπει να είναι γνωμοδότηση, κατά την άποψη της Επιτροπής μας, θα πρέπει να είναι μία γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Μεταφορών, γιατί κατά τη γνώμη μας ε, θα έπρεπε είναι, είναι τμήμα των αρμοδιοτήτων ε, της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ εφόσον η χρήση των ε, σαρωτών σώματος είναι κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με τις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης ε, επιτροπής, της Επιτροπής μας και το θέμα αυτό είναι και πολύ ευρύτερο από την ασφάλεια των αερομεταφορών μόνο. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι την πρώτη ε, την πρώτη φορά που ακούστηκε το θέμα των σαρατών ε, ε, σώματος υπόθηκε ότι κάποια στιγμή μπορεί να υποκαταστήσουν τους ανιχνευτές μετάλλων. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιείται πολύ περισσότερο από ό,τι μόνο στις αερομεταφορές. Οπότε νομίζω ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε περισσότερο τη λέξη σαρωτές σώματος και όχι σαρωτές ασφαλείας, ε, γιατί ε, ακριβώς ε, σαρώνει το σώμα του κάθε ατόμου. Δεν ξέρω, η Επιτροπή Μεταφορών χρησιμοποιεί περισσότερο την, την ε, έννοια σαρωτές ε, ασφαλείας. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα πρότυπα ασφαλείας για την χρήση των σαρωτών αυτών, δηλαδή να μην υπάρχουν ε, εικόνες πλήρης του σώματος, να μην αποθηκεύονται τα δεδομένα, να μην γίνεται επεξεργασία τους και Επίση, πρέπει να έχει κανεί τη δυνατότητα επιλογή να περάσει από το μηχάνημα αυτό ή όχι. Και αν επιλέξει να μην περάσει από το μηχάνημα αυτό, ε, πώ ε, θα του συμπεριφερθούν. Οπότε προφανώς ολόκληρη η διαδικασία ε, γύρω από το θέμα αυτό θα έπρεπε να συνάδει πλήρως με, το θέμα, με τα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδιωτικού βίου, προστασίας των δεδομένων και οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών είναι απαράδεκτη. Επίσης αναφέρθηκα και στο γεγονός ε, ότι οι σαρωτές που βασίζονται σε ε, ακτίνες χ ε, θα δεν θα μπορούσαν να είναι αποδεκτές γιατί αυτό διακινδυνεύει την υγεία των πολιτών και αν αυτό ε, αν θεωρείτε ότι είναι σημαντικό και απαράβατο δικαίωμα ε, η ασφάλεια είναι επίσης απαράβατο δικαίωμα το δικαίωμα του ανθρώπου να επιλέγει και γι' αυτό ε, πιστεύω ότι θα έπρεπε να ε, δούμε τι θα γίνει και με την Επιτροπή Περιβάλλοντος η οποία δεν απορρίπτει εντελώς την ιδέα των ακτίνων Χ. Θα έπρεπε λοιπόν να τους πούμε ε, καθαρά ότι εμείς δεν δεχόμαστε τις ακτίνες Χ και ότι αν το πούμε ευθαρσώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το ακούσει. Αν είμαστε λοιπόν πάρα πολύ σαφείς από αυτού ενδεχομένως ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει το ίδιο. Υπάρχει ένα ακόμη σημείο που θα ήθελα να επισημάνω που είναι το profiling. Η ισορροπία μεταξύ του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη καταπολέμηση τη τρομοκρατία, κατά την άποψη των πρασίνων, δεν θα έπρεπε να ακολουθεί ποτέ σε ε, πρακτικέ όπω το profiling. Και το λέω αυτό γιατί και στη γνωμοδότηση του ΕΜΒΗ υπάρχει μία πρόταση για profiling. Ε, Οπότε, αν κάνουν και εκείνοι ευρύτερε δηλώσει, θα κάνω και εγώ ευρύτερε δηλώσει στην Επιτροπή μα. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι η εισαγωγή των σαρωτών σώματος ενδεχομένω ή το γεγονός ότι ε, μπορεί και να μην εισαχθούν δεν θα έπρεπε ποτέ να οδηγήσει σε τέτοιου είδους πρακτικές. Θα ήθελα να ολοκληρώσω για την ώρα και θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σας ε, και να επανέλθω από αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σαρτζεντίνη. Είναι εδώ ο κύριος Κορνέλης, ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλετε να σχολιάσετε πριν αρχίσει η συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής μας. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Απλώς θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα να ενημερώσω τα μέλη της Επιτροπής σας για το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς αυτή τη στιγμή εκπονούμε τη μελέτη αξιολόγησης αντικτύπου που την είχαμε ανακοινώσει τον Ιούνιο του 2010. Είμαστε στα τελικά στάδια της ε, ε, μελέτης αυτής ε, και όταν θα ολοκληρωθεί θα ολοκληρωθεί δουλειά κατά αυτόν τον τρόπο και φυσικά επί τη βάση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενδεχομένως ε, να υπάρξει και μία πρόταση την οποία θα υποβάλουμε ε, μέσω της Επιτροπολογίας ε, κατά τους επόμενους μήνες. Τότε θα δημοσιευθεί και η μελέτη αξιολόγησης αντικτύπου και θα είναι διαθέσιμη σε όλους. Σας το λέω αυτό για να σας ενημερώσω ακριβώς που βρισκόμαστε από απόψεως εσωτερικής διαδικασίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κορνέλης. Μήπως ο κύριος Δεγκράντες ε, θα ήθελε τώρα να πάρει το λόγο. Γιατί θα αρχίσει η συζήτηση. Κύριε Δεγκράντες, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι η στιγμή να τοποθετηθώ και εγώ. Όπως είπατε είμαι σκιώδης εισηγητής ε, για το ΕΛΚ ε, και τη γνωμοδότηση της κυρίας Αργεντίνη και είμαι και εισηγητής επί της ε, για το θέμα αυτό στην Επιτροπή Μεταφορών. Θα ήθελα να πω, όσον αφορά την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, ότι δεν παρεμβαίνω ποτέ ε, όταν ε, υπάρχουν πολύ θεμητές, θεμητά αιτήματα από πλευράς της Επιτροπής αυτής. Όμως το είχα πει νομίζω και στην Ολομέλεια όταν, ε, τα, όταν πρόκειται για ένα ζήτημα θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, πρέπει να παρεμβαίνει η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Όμως, κύριε Πρόεδρε, ίσως θα έπρεπε να μην γνωμοδοτήσουμε πριν ε, δούμε την έκθεση, η οποία ακόμη μεταφράζεται. Για μένα, είναι μεγάλη τιμή να παρουσιάζω τη γνωμοδότηση αυτή ενώπιόν σας ως ε, αναπληρωματικό μέλος και νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσω να συζητήσω με την κυρία Σαρτζεντίνη για να δούμε κατά πόσο συμφωνούμε σε ό,τι αφορά τουλάχιστον ε, τις αρμοδιότητες ε, της Επιτροπής μας που πρέπει να ασχολείται με την πρόληψη και την υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το έχω πει άλλωστε και στην Επιτροπή Μεταφορών. Λόγω των ε, των τρομοκρατικών επιθέσεων δεν πρέπει να ασχολούμαστε μόνο με το θέμα των σαρωτών, πρέπει να ασχοληθούμε και με το θέμα των ε, υγρών γιατί όπως γνωρίζετε υπήρξαν και ε, κάποιες ε, απόπειρες επιθέσεων και σε αεροπορικές εταιρείες που μεταφέρουν ε, επιβάτες αλλά και σε εταιρείες που μεταφέρουν εμπορεύματα. Είναι και αυτό κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Είναι ένα ζήτημα λοιπόν που πρέπει οπωσδήποτε να το επιλύσουμε. Και θα ήθελα να πω το εξής. Το τελικό χτένισμα της έκθεσής μου το έκανα αφού, ε, αφού συμβουλεύτηκα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πολλές ομάδες εμπειρογνωμών και τις πολιτικές ομάδες σε σχέση με το κατά πόσο μπορούμε ή όχι να χρησιμοποιούμε τους συγκεκριμένους ερωτές. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε τους σαρωτές αυτούς, πρέπει να υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσει, ελάχιστες προδιαγραφές που να ισχύουν και μάλιστα οι απαιτήσει αυτές πρέπει να εφαρμόζονται ενιαία ώστε να μην υπάρχει σύγχυση ε, μεταξύ των επιβατών όπως ήδη ισχύει λόγω αυτής της κατάστασης. Οπότε, εγώ θα ήθελα να υποστηρίξω την έκθεσή μου, στην οποία λέω ότι τέτοιου είδους αρωτές πρέπει να είναι προαιρετικοί. Δηλαδή, ο επιβάτης αποφασίζει ναι ή όχι αν θα περάσει από το συγκεκριμένο σαρωτή και αν δεν θέλει να περάσει από το συγκεκριμένο σαρωτή, θα υποχρεούται ε, να υποβληθεί ε, σε ε, εξίσου αποτελεσματικούς ελέγχους, αλλά διαφορετικής φύσεως, ελέγχους που εξασφαλίζουν την ασφάλεια. Επομένως, το κράτος μέλος που χρησιμοποιεί τους συγκεκριμένους αρωτές πρέπει να σέβεται να τηρεί ορισμένους κανόνες ε, και ο επιβάτης αν δεν θέλει να περάσει από το συγκεκριμένο σαρωτή πρέπει να υποβληθεί σε άλλου είδους ελέγχους για να, να... να υπάρχει εγγύηση ασφάλειας για όλους τους υπολείπους. Σήμερα η Επιτροπή με πολύ καλές προθέσεις μας παρουσίασε ένα ε, πρόγραμμα για τους σαρωτές που δεν είχαν λάβει υπόψη ιδιαίτερες συνθήκες όπως για παράδειγμα τον ιδιωτικό βίο, την προστασία των δεδομένων, το σεβασμό των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και πρέπει η Επιτροπή να λάβει υπόψη την εντολή που της ε, δίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις επαφές μου με την ε, κυρία ε, Σαρτζεντίνη. Οι νέε τεχνολογίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ορίστηκαν σαφέστατα. Οπότε, Ποια είναι τα ζητήματα που μπορούν να μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Η προστασία δεδομένων, τα δεδομένα αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια του ελέγχου και στη συνέχεια πρέπει να καταστρέφονται. Τα δεδομένα αυτά δεν πρέπει να αποθηκεύονται, πρέπει να, να... να... να προστατεύεται επίσης ε... ε το ιδιωτική σφαίρα του, του κάθε ανθρώπου και μιλάω για τις εικόνες που παράγονται από τους συγκεκριμένους σαρωτές σώματος, όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να καταστρέφονται με συστηματικό τρόπο. Γιατί ε, υπήρξαν κάποιες, ε, ε, κάποια ε, πειράματα που έχουν αποδείξει ότι υπάρχουν άλλου είδους έλεγχοι που μπορούν σεβόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα να επιτύχουν το ίδιο επίπεδο ασφάλεια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να διαλέξει το ένα ή το άλλο σύστημα. Εγώ δεν πρόκειται να κάνω κάτι τέτοιο στην έκθεσή μου. Δεν θα πω ότι το ένα σύστημα είναι καλύτερο από το άλλο. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να γίνεται με κάποια διακριτικότητα και υπάρχουν κάποιες άλλες λεπτομέρειες που δεν πρέπει να γίνονται γνωστές ε, σε σχέση τώρα με αυτά που μας είπε η κυρία Σαρτζεντίνη και την δική της άποψη, πρέπει να πω ότι όντως μπορώ να συμφωνήσω με μερικά από τα σημεία που επεσήμανε, όμως υπάρχει και μία διαφορά που θα ήθελα να τονίσω είναι θεμητό η, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών να ασχολείται με ε, την, ε, ε, τους κανονισμούς που αφορούν τους σαρωτές σώματος και τις πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. και ότι αυτό δεν αφορά μόνο τις αεροπορικές εταιρείες. Πρέπει ε, τις αεροπορικές μεταφορές. Μερικές φορές μπορεί να χρησιμοποιηθούν για παράδειγμα στα μουσεία. Και δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να αποστείλουμε ένα τέτοιο είδους μήνυμα. Είναι λίγο ευαίσθητο το ζήτημα αυτό και με το σχόλιο αυτό θα ολοκληρώσω και την παρουσίασή μου για να μην βαρεθείτε. Στην έκθεσή μου συμφωνώ ο στην έκθεσή μου αναφέρω ότι συμφωνώ ότι η ακτίνες χ δεν είναι πάντοτε εναλλακτική λύση. Πρέπει τις ε, ε, έγκυες γυναίκες, τα παιδιά, ε, τα, τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού να τις προστατεύσουμε από τις επιβλαβείς συνέπειες των ακτίνων χ. Επομένως οι ακτίνες χ πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν αυτό επιτρέπεται και να απορρίπτονται στο πλαίσιο των ε, ε, σαρωτών σώματος. Τα κράτη-μέλη βέβαια έχουν το δικαίωμα που δεν μπορεί να τους το αφαιρέσει κανείς να επιβάλλουν αυστηρότερα μέτρα από τα μέτρα που θα αποφασίσουμε εμείς και με αυτό θα θέλω να ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται λοιπόν για ένα θέμα για το οποίο δεν συμφωνώ απολύτως με την κυρία Σαρτζεντίνη. Και θα διαβάσετε την έκθεσή μου, θα τα δείτε άλλωστε όλα αυτά. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε την ε, δυνατότητα να ακούσουμε και την κυρία Σαρτζεντίνη, αλλά προηγουμένως θα ακούσουμε τα μέλη της Επιτροπής που ήθελαν ε, να παρέμβουν στη συζήτηση. Ο κύριος Σουμπούτη, ε, όχι, έχουν ε, αναφερθεί τα σχόλια μου, καλύφθηκα. Ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, χαίρομαι που ε, επιτέλους συζητούμε αυτή την έκθεση. Αφιερώσαμε πολύ χρόνο να να στη συζήτηση του αν το άρθρο 50 ή όχι. Αλλά η Επιτροπή Μεταφορών ζήτησε ε, καταρχάς αυτή την ε, ε, έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Και υπήρχαν τόσα πολλά θέματα που αφορούν τις αερομεταφορές που εμπίπτουν στις δικές μας δικαιοδοσίες που θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να έχουμε και εμείς λόγο. Ε, είπαμε στην Επιτροπή Μεταφορών ότι το θέμα των σαρωτών σώματος είναι πάρα πολύ επίκαιρο και νομίζω ότι στην Επιτροπή ΛΥΠΕ σε αυτό συμφωνούν όλες οι πολιτικές ομάδες. Ε, υπάρχει ζήτημα θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως είναι το profiling, η απεικόνιση του σώματος και ε, η έμφυλη απεικόνιση του σώματος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλει να κάνει η Επιτροπή μας, αυτό που θέλει να κάνει η κυρία Σαρτζεντίνη, είναι να συμβάλλουμε όσο γίνεται πιο επικοδομητικά στην έκθεσή σας ελπίζουμε να δούμε αυτή την έκθεση γιατί μόνο τότε θα μπορέσουμε να αναλύσουμε το βασικό ζήτημα που είναι το εξής, ότι οι σαρωτές σώματος έχουν μια πολύ δύσκολη ιστορία πίσω τους. Ε, είχα την ευκαιρία να δω την τεχνολογία αυτή στην πράξη σε δύο ε, αεροδρόμια ε, στο Μάντσεστερ, ίσως το ξέρετε κι εσείς, και η κυρία Σαρτζεντίνη, αλλά και στο Χήθρο, όπου γίνονται κάποιοι τέτοια έλεγχοι. Το θέμα των θελμιωδών δικαιωμάτων για μας δεν είναι το κατά πόσο είναι εθελοντικό το πέρασμα από του ερωτές ή όχι. Νομίζω ότι και εσείς και η κυρία Σαρτζεντίνη συμφωνείτε ότι θα πρέπει να είναι εθελοντικό το κατά πόσο θα περνάει κανεί από αυτού του ερωτές ή όχι. Το πραγματικό πρόβλημα όμως που έχουμε είναι πρώτα απ' όλο ότι υπάρχει ε, διαφορά μεταξύ των διαφόρων αεροδρομίων, ε, πράγμα το οποίο δημιουργεί σύγχυση στο κοινό που ταξιδεύει και δεύτερον ε, είναι το κατά πόσο χρησιμοποιούνται ίδιου είδους σαρωτές στα μεγάλα αεροδρόμια. Έχω δει διάφορες εικόνες και όλες οι εικόνες που έχω δει δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι ε, ε, δείχνουν ότι υπάρχει ένας υπάλληλο, ένα ξεχωριστό παραβάνασμα που κάθεται και βλέπει την εικόνα που παράγεται ε, για να δει αν υπάρχει κάτι το επικίνδυνο. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε και το περίγραμμα του ανθρώπινου σώματος έτσι. Και θέλω να δω για το θέμα αυτό την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών για να δούμε ποιο είναι το νόημα της χρήση αυτής της τεχνολογίας. Το κατά πόσον όλοι οι σαρωτές σώματο δείχνουν τέτοιου είδους εικόνες. Διότι η κυρία Σαρτζεντίνη ε, γράφει στην έκθεσή της ότι θα έπρεπε να δημιουργούνται ένα είδους ε, ανώνυμες ε, εικόνες, ομοιόμορφες εικόνες. Δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο ισχύει, διότι υπάρχει θέμα ιδιωτικής ζωής ε, και οι εικόνες αυτές πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, έχετε ακούσει φαντάζομαι ότι κάποιες αυτές τις εικόνες έχουν διαρρεύσει και βρίσκονται τώρα στο διαδίκτυο. Το δεύτερο ζήτημα είναι το θέμα του profiling και άλλα θέματα ασφαλείας που σχετίζονται μεταξύ τους. Και θα πρότεινα στη συνάδελφο την Τζούντιθ Σαρτζεντίνη να κάνει κάποιες τροπολογίες στη γνωμοδότησή της που να αφορούν και κάποιους άλλους τομείς της ε, ε, ασφάλειας γιατί οι σαρωτές σώματος δεν φαίνεται να είναι το μόνο ζήτημα που υπάρχει σε σχέση με την ασφάλεια. Και τέλος, θέλω να πω ότι θα έπρεπε να συνεργαστούμε πολύ στενά, γιατί η ταχύτητα με την οποία ε, δοκιμάζεται αυτή η τεχνολογία και η ταχύτητα με την οποία τα διάφορα μεγάλα αεροδρόμια αλλάζουν την πολιτική τους δημιουργεί τεράστια σύγχυση. Ε, και στην έκθεσή σας, στη δική σας, της Επιτροπής Μεταφορών, θα έπρεπε ε, να υπάρχει κάποια αναφορά στο θέμα αυτό. Γιατί τα πράγματα κινούνται πάρα πολύ γρήγορα, η τεχνολογία κινείται ραγδαία. Όλοι θέλουμε να είμαστε προστατευμένοι, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να προκύψει μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λέει στην κοινή γνώμη πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει μεγάλη σύγχυση. Ε, τα διάφορα μεγάλα αεροδρόμια δημιουργούν, χρησιμοποιούν το καθένα διαφορετικά συστήματα ασφάλειας ε, και διαφορετικούς αρωτές. Ε, είναι πραγματικά λοιπόν πολύ δύσκολο ε, να συλλάβουμε τον πυρήνα του προβλήματος η συζήτηση αναφίβολα θα είναι ενδιαφέρουσα. Περιμένουμε να δούμε την ε, έκθεσή σας και θα υποβάλουμε για κάποιες τροπολογίες τη γνωμοδότηση της κυρίας Αργεντίνη. Ευχαριστώ. Κυρία Νετφέλτ, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστώ και τους δύο συγκητές για τη δουλειά τους και να πω ότι σε μεγάλο βαθμό συμμερίζομαι την προσέγγιση κυρίας Αργεντίνη. Η ομάδα μου όμω. προτίθεται να καταθέσει μια σειρά τροπολογιών με στόχο όχι τόσο να τροποποιήσει το κείμενο όσο να το συμπληρώσει με κάποια στοιχεία. Πρώτον, και δεν αναφέρομαι σε τροπολογία, αλλά σε πιο γενικό ζήτημα, το ζήτημα της αρμοδιότητας, ποια, ποια επιτροπή είναι αρμόδια. Επειδή μιλάμε για σαρωτέ σώματο σε αεροδρόμια, παίρνει το θέμα στην αρμοδιότητα τη Επιτροπή των Μεταφορών. Εάν όμω, από, ό,τι φαίνεται αυτό ισχύει, μιλούμε για στρατό σώματο οπουδήποτε αλλού, δεν υπάρχει λόγο να υπαχθεί στι ε, μεταφορέ το θέμα αυτό. Είναι νομικό ζήτημα καθαρά και άρα θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά, πιστεύω. Γιατί είναι ένα ζήτημα που, όπω είπε και ο Κλωτ Μωρέ, ε, απέτειται των ε, ζητημάτων τη ασφάλεια και των πολιτικών ελευθεριών. Δεύτερον, Θα θέλω να επισημάνω ότι διαρκώ δεν πρότεινα το ίδιο σφάλμα. Δηλαδή, μπαίνουμε, πέφτουμε στην παγίδα τη συζήτηση των λεπτομεριών, χωρί να διαρωτηθούμε αν πράγματι χρειάζεται κάτι τέτοιο. Ή να ορίσουμε τι προσδοκίε έχουμε. Έχουμε ορίσει ποιε είναι οι προσδοκίε μα. Όχι από ό,τι φαίνεται. προσδοκία μας τι είναι, να συλλάβουμε κάποιον τρο, επίδοξο τρομοκράτη ο οποίος θέλει να μπει μέσα σε ένα αεροπλάνο, σε ένα εμπορικό κέντρο φορτωμένος με ε, εκρηκτικά. Γιατί αν είναι έτσι, δεν πρόκειται να μας βοηθήσουν αυτοί οι σαρωτέ γιατί αν είναι κρυμμένα μέσα σε κοιλότητες του σώματος τα εκρηκτικά, δεν τα βλέπει ο σαρωτή σώματος, Άρα, τι εξυπηρετεί ακριβώς. Ε, ε θέλουμε να συλλάβουμε άλλου τύπου ε, εγκληματικές δραστηριότητες, φερρυπίν ε, λαθρεμπόριων ναρκωτικών. Εκεί ναι, μπορεί να έχει νόημα να καταπολεμήσουμε το λαθρεμπόριο των ναρκωτικών, αλλά άλλο είναι να, να προσπαθούμε να προλάβουμε έναν επίδοξο τρομοκράτη και άλλο είναι να προσπαθούμε να συλλάβουμε κάποιο λαθρέμπορο ναρκωτικών. Πρέπει να υπάρχει και ένα μέτρο. Αυτό νομίζω λοιπόν ότι λείπει, ότι δεν έχουμε προσδιορίσει σαφώ στόχου. Και αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που το παθαίνουμε. Δεύτερον, ένα άλλο ζήτημα που παραβλέπουμε συνήθως είναι το οικονομικό. Όταν έγινε η πρώτη συζήτηση μεταξύ της Επιτροπής Μεταφορών και, Πολιτικών, και της ε, Επιτροπής των Πολιτικών Ευθυριών, πρέπει να ακούσω κάποια ε, ε, αιτιολόγηση πλευρά Ευρωπαίκη Επιτροπής, να πει δηλαδή ότι κάποια κράτη-μέλη διανοούνται τη θέσπιση έστω και υποχρεωτικά ακόμη αυτών των σαρωτών και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να έχουμε μια συλλογική προσέγγιση όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα το οποίο εκ πρώτης όψης φαίνεται λογικό. Εάν όμως η Επιτροπή μας λέει ότι ορισμένα κράτη έχουν προχωρήσει σε πιλωτικές δοκιμές, τι οποίε όμω έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι σαν να είμαστε σε ένα ασφάβολο κύκλο στην επιχειρηματολογία μας Χρειάζεται λοιπόν απόλυτη διαφάνεια. Ποιο έχει χρηματοδοτήσει αυτά τα πιλωτικά σχέδια, τι δοκιμέ, ποιο θα χρηματοδοτήσει την εγκατάσταση των σαρωτών και χρειάζεται απόλυτη διαφάνεια για το κόστο. Γιατί τίνουμε εδώ στο Κοινοβούλιο να εγκρίνουμε νομοθεσία χωρί να γνωρίζουμε ποτέ πόσο θα μα κοστίσει. Και στην ελευθερία και πόσο αξίζει αυτή την οικονομική επιβάρυνση. Δεν νομίζω να υπάρχει Εθνικό Κοινοβούλιο το οποίο να τολμά να εγκρίνει νομοθεσία χωρί τελικά να ξέρει τι λογαριασμό θα κληθεί να πληρώσει ο φορολογούμενος. Μπα περιπτώσει ξέρουμε ότι θα υπάρχουν δημοσιονομικέ ε, συνέπειε και θέλουμε να είναι σαφή η εικόνα πριν να εγκρίνουμε αυτών των οικονομικών συνοπιών. Επίση, ε, θελοντική ή μη υπαγωγή στον έλεγχο. Τι σημαίνει θελοντική. Ε, το εθελοντική υπαγωγή τι σημαίνει, αν κάποιος αρνηθεί να περάσει από τον ε, έλεγχο αυτού του σαρωτή, ε, χωρίς να θέλω να σας περιγράψω τις φρικτές λεπτομέρειες, τουλάχιστον στις Πολιτείες ε, υφίσταται έναν διεξοδικό, όπως ονομάζεται, ε, σωματικό έλεγχο, που είμαι σίγουρη ότι θα σας είναι ευχάριστος. Και είναι πολλοί αυτοί στις ΗΠΑ οι οποίοι αντιδρούν. Εναλλακτική δηλαδή δεν υπάρχει είμαστε υποχρεωμένοι περισσότερο να περάσουμε από τον έλεγχο αυτών. Επίσης υπάρχει εμπειρία στις Πολιτείες και καταχρήσεις υπάρχουν γιατί ο κόσμος μας δεν είναι ιδιώδης. Υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι αποθηκεύουν τις φωτογραφίες και μετά αυτές διαραίουν. Υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι φτιάχνονται να βλέπουν τις εικόνες ε, μέσα από το σαρωτή ανθρώπων του άλλου φίλου ή και του ίδιου φίλου ακόμη. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν οι διάφοροι ανώμαλοι, υπάρχουν οι διάφορες ε, καταχρήσεις και θα πρέπει να υπάρξουν αυστηρότατες ποινές, ακόμη και φυλάκιση για οποιονδήποτε καταχράται αυτή τη χρήση του ε, Και τελική παρατήρηση. στην πατρίδα μου και φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη η κυβέρνησή μας αρνείται να δώσει πλήρε πληροφορίες για τις τεχνικές, για τα τεχνικά στοιχεία του ε, Σαρωτή. Ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες που έγινε σχετική μελέτη από το Κογκρέσο απεδείχθη ότι Υπάρχει ε, παραγγελία από την Αμερικανική κυβέρνηση ενός αρωτή ο οποίος έχει τη δυνατότητα και να αποθηκεύσει και να ε, παραγάγει, να αναπαραγάγει μάλλον την εικόνα. Πράγμα το οποίο είχε δεσμευθεί η Αμερικανική κυβέρνηση όταν το έπρεπε. Γιατί λοιπόν έχω να πιστέψω ε, την κυβέρνησή μου ότι δεν πρόκειται να κάνει το ίδιο πράγμα. Παρά ό,τι σας διαβεβαιώσει μπορεί να μου δώσει. Εδώ νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με ένα σοβαρό ζήτημα και αν, και αν συμφωνεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει ε, με το νόμο του Δούνε και Λαβίνη λίγο πολύ να διεκδικήσουμε να έχουμε μια πλήρη, πλήρη ε, επισκόπηση των τεχνικών στοιχείων. Ευχαριστώ κύριο πρώτα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως ξέρετε πρόεδρε, Έχω πολύ αγωνιστεί για το θέμα που έχει να κάνει με την αρμόδια της ουσίας επιτροπή και για τα όσα είπε και ο Κλώτ συμφωνώ ότι έχουμε συμφωνήσει, έχουμε συζητήσει μάλλον επί μακρόν το γεγονός ότι θα πρέπει την αρμοδιότητα να την αναλάβει η δική μας επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει όμως τουλάχιστον μπορώ να έχω την ικανοποίηση ότι έχουμε δύο εξαίρετους ε, εισηγητές, τον κύριο Λουίς Δεγράντε, μας εκπροσωπεί στην αρμόδια κατ' επιτροπή και την κυρία Σαρτζεντίνη. Για τη γνωμοδότηση. Κάποια ζητήματα λοιπόν τώρα. Μέχρι τώρα δεν είχαμε την ευκαιρία, τη δυνατότητα να διαβάσουμε το όσα γράφουν οι εισηγητές. Μπορεί να ακούσαμε τι χαρά μας αλλά δεν τα διαβάσαμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες ιδέες, οι οποίες δεν ήθελα να συμπληρώσω ή να τοποθετηθώ, για να διευκρινίσω κάποια ζητήματα. Φερρυπίν. Έκθεση τέτοιου τύπου θα πρέπει να υπάγεται σε τέσσερις προϋποθέσεις. Νομικά, καταρχάς το κριτήριο της αναλογικότητας, αλλά και της επικουρικότητας, όπως και των οικονομικών συνεπειών. Δεύτερον, Μιλάμε για την ασφάλεια των ενέργειων μεταφορών συγκεκριμένα, όχι των οδικών, όχι των θαλασσίων, ούτε των ε, άλλων ε, πλωτών οδών, ποταμών κτλ. Μιλούμε λοιπόν για ενέργειες μεταφορές και για σαρωτές σώματος. Για να δούμε λοιπόν. Για να Τι θέτε εδώ ζήτημα εναρμόνισης, από ό,τι φαίνεται το έχουν ξεκαθαρίσει και οι κάποιων αξιών που είναι οι εξή πολύ απλά. Της υγείας, της προστασίας των ε, προσωπικών δεδομένων, της προσωπικής, του προσωπικού βίου, της αρχής αναλογικότητας με την ελάχιστη δηλαδή ε, ζημία για τον εμπλεκόμενο και της καταστροφής σε πραγματικό χρόνο των εικόνων. Αυτή είναι βασικά η, η ουσία πάνω στην οποία εργαζόμαστε. Και πρέπει βέβαια στις δύο εκθέσεις να συμπεριλαμβάνουν τέσσερις ε, βασικές αρχές, η οποίες Πρώτον, η αποτροπή. Τη λέξη αποτροπή δεν την άκουσα πουθενά. Είναι ουσιώδου σημασία η λέξη αποτροπή. Η πρόληψη, δεύτερον, τρίτον, και δεν είναι το ίδιο με την αποτροπή, τρίτον, διάγνωση, ανείχνευση καλύτερα, και τέταρτον, προστασία ή σεβασμός μάλλον των θεμελιδών δικαιωμάτων στο επόμενο επιχείρημα. Η απόφαση θα είναι απόφαση των ελάχιστων κοινών προνομαστή, όπω πάντα όταν λαμβάνουμε αποφάσει ε, για τα 27 κράτη-μέλη. Υποχρεωτική λοιπόν ε, διέλευση για του επιβάτε. Πολύ καλά. Όλοι όμω γνωρίζουν ότι αν ο επιβάτη αρνηθεί να περάσει από αυτά τα φίλτρα ασφαλεία, θα τον υποβάλει ή θα επιβάλλει καλύτερα με βάση την αρχή της επικουρικότητας στο κράτος ε, μέλος ε, κάποιους εναλλακτικούς ελέγχους ε, που θα είναι έλεγχοι σωματικοί, πολύ πιο περίπλοκοι και ως προς τα θέματα της υγείας των ανθρωπινών δικαιωμάτων και το καθεξής. Άρα είναι μια υπόθεση αυτή πολύ δύσκολη, λεπτή και θα πρέπει να την εξετάσουμε και υπό την έννοια της αρχής του de Επίσης θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε ή να καθασίσουμε σαφέ μέσα στι εκθέσει το τι είναι σωματικός σαρωτής, σαρωτής σώματος δηλαδή για τις εναέριες ε, μεταφορές και τι είναι ο σαρωτής ασφαλεία, γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα Άλλο είναι, άλλη δουλειά κάνει ο καθένας και δεν μπορεί πάντοτε να διαγνώσει την μεταφορά παράνομων ουσιών ή, ή εκρηκτικών. Αυτές οι παρατηρήσεις είχα. Πιστεύω ότι με αυτά ε, θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τους ε, δύο εισηγητές μας ε, σε αυτό το δύσκολο έργο που έχουν αναλάβει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σίπελ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια πολύ απλή ερώτηση. Το αν προσπαθούμε με την αλλαγή μιας λεξούλας εδώ και εκεί να χαράξουμε πολιτική. Πού, ποιος είχε την ιδέα ότι μιλάμε για σαρωτές ασφαλείας. Για να μιλάμε για σαρωτές ασφαλείας πρέπει να έχουμε μία, μάλλον η ασφάλεια για να το πω έτσι, πρέπει να ε, ε, εκπροσωπείται με ένα υλικό αντικείμενο, με ένα αντικείμενο που πρέπει να πιάσει και να δει. Αυτό δεν υπάρχει λοιπόν. Αυτό λοιπόν μόνο καλύπτεται μέσα από τις εκθέσεις μέσα από τις τοποθετήσεις κατά αυτών των ε, σκάνερ σώματος, ερωτών σώματος, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι προβλήματα γεννούν, όχι μόνο προς την ε, προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά το κατά πόσον μπορούν να ε, αποθηκευτούν οι εικόνες, ακόμη και αν δεν φαίνονται στην οθόνη, και σε ποιο βαθμό μπορούν να εξαχθούν από αυτού του ερωτέ οι εικόνε, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και στη τελευταία ανάλυση το κύριο ερώτημα είναι σε τι κερδίζουμε σε περισσότερη ασφάλεια χάρη σε αυτού του ερωτέ. Αυτή την απάντηση δεν έχουμε λάβει ακόμα. Και εγώ πιστεύω ότι αυτή η νέα ιδέα του σαρωτή ασφαλείας είναι απλώς στάχτη στα μάτια όποιων δεν γνωρίζουν τα πράγματα αρκετά καλά, ε, για να ε, αποτρέψουν την υποβολή οποιονδήποτε ερωτήσεων από εκείνους που δεν έχουν μελετήσει καλά την υπόθεση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει σε ερωτήσει ασφαλείας, δεν προσφέρει προστηρία ασφάλεια και πρέπει να κάνουμε ένα ανοιχτό διάλογο, δημόσιο διάλογο με την κοινή γνώμη για το τι είδους ασφάλεια θέλουμε, με ποιο τίμημα και με τι επιπτώσει για την ε, ανθρώπινη εξωτερική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Μποσκούρτ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και τους δύο εισηγητάς, οι συντάκτες καλύτερα. Και η κυρία Σαρζεντίνη έχει διάφορα θέματα προτείνει να κτιστείς και για τον κύριο Ντεγκράτας Πασκουάλ θα ήθελα να ποσο κάποιες ερωτήσεις γιατί λέτε ότι ο σαρωτής σώματος θα πρέπει για να εισαχθεί να ε, εγκρίνεται από το κάθε κράτος μέλος χωριστά, αν κατάλαβα καλά. Δηλαδή να υπάρχουν μόνο ελάχιστες προδιαγραφές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην το αποφασίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό είναι ο τρόπος να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Μήπως τελικά δηλαδή κάποιος προτιμάει μετά να μεταβεί, να ταξιδέψει σε ενός αεροδρομίου που δεν διαθέτει σαρωτισώματος. Για δε την υγεία του ανθρώπου, τι συνέπειες μπορεί να έχουν αυτοί οι σαρωτές. Δεν είναι καθόλου ξεκάθαρη η κατάσταση, κυρία Πασκουάλ. Και ακόμη μια ερώτηση σε σχέση με τις εναλλακτικέ που ενδεχομένω προτείνονται. Εάν δεν υπάρχει δηλαδή πρόθεση, αν δεν θέλει ο ταξιδιώτης να περάσει μέσα από τον σαρωτή σώματος, τι συνέπειες μπορεί να υπάρχουν. Γιατί δεν νομίζω να χαίρεται κανείς να περάσει μέσα από το μηχάνημα. Δηλαδή μπαίνει κανεί στο μηχάνημα, βλέπει ένα κόκκινο φως το οποίο τον ε, διαπερνάει από πάνω μέχρι κάτω Λέτε ότι εναλλακτικά, το είπε η κυρία Νετφέλτ, υπάρχουν άλλες λύσεις σωματικού, ε, σωματικής έρευνας. Συγκεκριμένα λοιπόν τι εννοείτε. Παρακαλώ. Κυρία Αλφάνο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ απολύτως με όσα είπαν μέχρι τώρα οι συνάδελφοι. Το να αντιμετωπίσουμε το θέμα των σαρωτών σώματος είναι ε, ζήτημα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και πρέπει να ξαναδούμε επίση σε σχέση με αυτό και το θέμα των υγρών που επιτρέπεται να μεταφέρονται σε σχέση με αυτήν την οδηγία. Όμω, ε, η παράγραφος 3 φαίνεται ότι οδηγεί σε λανθασμένες ερμηνείες που σίγουρα δεν είναι η πρόθεση της ε, εισηγήτριας. Φαίνεται να θέλει να ρυθμίσει το θέμα της χρήσης των σαρωτών σώματος και εκτός των αεροδρομίων ε, ειλικρινά ε, δεν είναι αυτή η πρόθεση. Μετά έχω μία ερώτηση για την ε, Κομισιόν. Και η δική μου χώρα εγκατέλειψε σχεδόν παντελώς τη χρήση των σαρωτών σώματος. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, πόσα είναι τα κράτη-μέλη που χρησιμοποιούν αυτούς τους σαρωτές και σε σχέση με αυτόν τον αριθμό, αν είναι απαραίτητο τελικά να ε, ρυθμιστεί η χρήση αυτών των μηχανημάτων για τα οποία από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχει ακόμα καμία βεβαιότητα. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω κατά προσέγγιση όσο δυνατόν ε, πιο ακριβή ε, ποιος είναι ο αριθμός, είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός των κρατών μελών που χρησιμοποιούν ήδη αυτόν τον εξοπλισμό. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι κάναμε μια συζήτηση εμπεριστατωμένη. Νομίζω ότι θα ακούσουμε την εισηγήτρια της ε, Επιτροπής μας, την κυρία Σαρτζεντίνη, αλλά προηγουμένως ίσως θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε λίγα λεπτά για να δοθεί μια απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση που έκανε η κυρία Αλφάνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το πόσο χρησιμοποιούνται οι σαρωτές σώματος στην Ευρώπη. Η Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με πληροφορίες ε, εξακολουθεί να υπάρχει απειλή για την πολιτική αεροπορία και αυτό είναι ο λόγος ε, για τον οποίο εργαζόμαστε επί του ζητήματος αυτού. Επίσης, ε, έχουμε πολύ λεπτομερή νομοθεσία για τις αερομεταφορές που δεν έχουμε σε άλλους τομείς και αυτό μας επιβάλλει να το εξετάσουμε πολύ προσεκτικά και να είναι τμήμα του προγράμματό μα. Γι' αυτό ακριβώ θέλουμε να το δούμε ε, το θέμα αυτό συγκεκριμένα για το θέμα των αεροπορικών μεταφορών. Επίσης, ε, πολύ σωστά υπενθυμίσατε την, ε, το ιστορικό της όλης πρότασης. Πριν από κάποια χρόνια είχαμε συζητήσει τους αρωτές σώματος ως ε, δυνατότητα σάρωσης χωρίς να βλέπουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες του ανθρώπινου σώματος και από τότε εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να δούμε όλες τις πτυχές από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ζητήσαμε επίσης καθοδήγηση και κάναμε και δημόσια δημόσια Και όπω είπα και προηγουμένω, βρισκόμαστε και στα τελικά στάδια τη μελέτη αξιολόγηση αντικτύπου, που εξετάζει όλε τι πιθανέ συνέπειε των σαρωτών ε, σώματος, κοινωνικά, οικονομικά ζητήματα, ζητήματα ε, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, είναι λοιπόν όλα αυτά θέματα που μας απασχολούν και τα εξετάσαμε εις βάθος και πρόκειται για θέματα τα οποία και εσείς αναφέρατε στην συζήτηση, στη συζήτηση σήμερα. Το πρώτο θέμα που προέγυψε πριν από μερικά χρόνια είναι από τη μία ήδη υπάρχουν ε, πολλές τεχνολογικές πρόοδοι και πρόκειται άλλωστε για έναν τομέα με πολλές ε, τεχνολογικές εξελίξεις που μας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι μηχανές από μόνες τους είναι τέλειες ε, και ε, θέλουμε βέβαια να υπάρχουν κάποιες εγγυήσεις, κάποιες συνθήκες λειτουργίας των συγκεκριμένων μηχανημάτων και φυσικά και χρήση των σαρωτών αυτών. Για ορισμένα συγκεκριμένα ζητήματα που ετέθησαν, μία ερώτηση αφορούσε την τεχνολογία για τα stick figures, stick figures δηλαδή το περίγραμμα του σώματος χωρίς ε, ε, ε καταγραφή, χωρίς εμφάνιση φύλου ε, εμάς, εμείς θα διστάζαμε ε, για πολύ λεπτομερή ρύθμιση της τεχνολογίας ε, γιατί ουσιαστικά έτσι ευνοούμε έναν συγκεκριμένο παραγωγό αν είμαστε πάρα πολύ, συγκεκριμένο κατασκευαστή αν είμαστε πάρα πολύ λεπτομερείς γι' αυτό προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ουδέτεροι από απόψεις της τεχνολογίας αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε και γενικές συνθήκες χρήσης των μηχανημάτων δεν ε, θέλουμε κανένα είδους profiling ε, στο πλαίσιο του θέματος αυτού των σαρωτών και όσον αφορά τη χρηματοδότηση μπορώ να σας ενημερώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει χρηματοδοτήσει κανένα πιλωτικό πρόγραμμα για τους ε, σαρωτές ε, ούτε δοκιμές, ε, άλλωστε δεν θα είχαμε και τον προπολογισμό να το κάνουμε, ακόμη και να το θέλαμε. Αυτό γίνεται από τα κράτη-μέλη και είναι τμήμα ε, της νομοθεσία μας. Τα πιλωτικά προγράμματα και οι δοκιμές ενθαρρύνονται, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να ξέρουμε για τι, τίποτε για τις χρήσει και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. Ε, και άλλωστε έχει εξελιχθεί και η τεχνολογία ακριβώς επειδή υπήρξαν πιλωτικά προγράμματα και δοκιμές. Όσον αφορά τώρα το κόστος, θα καλύπτεται το θέμα των σαρωτών ε, στις, και κατά πόσο θα καλύπτεται το θέμα αυτό ε, στην μελέτη αξιολόγηση αντικτύπου. Ναι, θα καλύπτεται. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, η Δανία ε, έχουν προβεί σε πιλωτικά προγράμματα και σε δοκιμές για τη χρήση των σαρωτών σώματος και η Γερμανία ε, και επίσης σε δοκιμές έχουν προβεί και η Γαλλία και η Ιταλία. Αλλά βέβαια δεν είναι μία επιτρεπόμενη για την ώρα μέθοδος ελέγχου. Οπότε μπορούν μόνο σε δοκιμαστική βάση να χρησιμοποιούν τα μηχανήματα αυτά ε, στα συγκεκριμένα κρατημέλη που ανέφερα. Ελπίζω να ανακάλυψε τα περισσότερα ερωτήματα. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σαρτζεντίνη, για το τελικό σχόλιο. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις και πολλές παρατηρήσεις. Βλέπω ότι κοιτάτε και το σκιώδη συγητή μας. Ε, ε στην ΛΥΜΠΕ και θα προσπαθήσω να καλύψω τα βασικότερα ερωτήματα, όπω και το ερώτημα τη κυρία Πόσκορτ για παράδειγμα, προ τον κύριο Ντεγκράντε Πασκουάλ. Καταρχά, αν χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε τέτοιου είδου μηχανήματα που έθεσε η κυρία Ίνετφελτ, Κοιτάξτε, ε, τα, ε, έχουμε ελάχιστε προδιαγραφέ αυτή τη στιγμή. Ε, Αυτέ θέλουμε να επιτύχουμε. Δεν θα ήθελα να σα απαντήσω λοιπόν πλήρω αν τα χρειαζόμαστε ή όχι τα μηχανήματα αυτά. Μάλλον θα χρειαζόμαστε αν πρέπει να σας απαντήσω και όχι γιατί είναι δική μου πεποίθηση αλλά γιατί είναι η άποψη πλειοψηφίας. Αμφιβάλλω όμως, οπότε θέλω ελάχιστες προδιαγραφές. Αυτό προσπαθώ να επιτύχω. Αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε είναι μέσα καταπολέμησης της ε, τρομοκρατίας. Ε, όποιος λοιπόν είναι αφοσιωμένος στην καταπολέμηση του εγκλήματος, ε, δεν θα πρέπει να το ε, ε μαζί με αυτό το θέμα γιατί νομίζω ότι έχουμε αρχίσει ήδη να κάνουμε κατάχρηση ενός μηχανισμού για λάθος λόγους. Ο κύριος Δεγκράντες που είναι και εισηγητής στην Επιτροπή Μεταφορών το κατέστησε σαφές και χαίρομαι ιδιαίτερος ότι θα πρέπει να είναι εθελοντική η χρήση Καταλαβαίνω τις ε, παρατηρήσεις ε, των συναδέλφων για το τι είναι, τι θα πει εθελοντική χρήση. Αν όμως οι προδιαγραφές μας είναι ορθές, ενδεχομένως να μην υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Ε, αλλά αυτό εξαρτάται από τις ελάχιστες προδιαγραφές. Και νομίζω και την ερώτηση του κυρίου Μωράης απαντά αυτό, που ανέφερε τις κυρώσεις για την, για την κατάχρηση. Ε, ναι, το γνωρίζω τον αεροδρόμιο του Μάντσεστερ. Είναι το χειρότερο παράδειγμα που μπορείτε να δώσετε. Στο Χίθρο, για παράδειγμα, κάποιο να κάθεται και να βλέπει φωτογραφίε από απόσταση, δεν νομίζω ότι αυτό είναι τμήμα ελαχίστων προδιαγραφών. Και η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή είπε επίση ότι θα ήθελε μια ε, ε, ουδέτερη τεχνολογία και το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ δεν να μην το κάνουμε αυτό, απλώς λέω να έχουμε την πιο προηγμένη τεχνολογία και να έχουμε ελάχιστε προδιαγραφές ορχε, ε, ορθές. Και γι' αυτό νομίζω σε σχέση με τις ακτίνες χ ότι δεν θα πρέπει να λέμε τι είδου σαρωτή θα έχουμε, αλλά πρέπει να είναι σαφέ τι είδου μηχάνημα δεν πρέπει να έχουμε. Εγώ δεν είμαι στην Επιτροπή Μεταφορών, τώρα είμαστε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, αλλά φανταστείτε ότι κάποια αεροδρόμια έχουν ακτίνε χ και κάποια άλλα αεροδρόμια έχουν κάτι άλλο. Εγώ πως επιβάτη, πώς θα γνωρίζω κατά πόσο είναι ασφαλέ το ένα ή το άλλο μηχάνημα και φανταστείτε τι θα γίνει αν αυτή που λέει, αν, η, μια γυναίκα λέει ας πούμε ότι είναι έγκυος, ε, οι πιλότοι, παιδιά, ε, δεν θέλουν να περάσουν από, τις, ε, από τους αρωτές γιατί θεωρούν ότι έχουν ακτινισχύ. Α, δεν μπορούμε να πούμε εμείς στις περιφέρειές μας καλούτσικο είναι ή χαμηλή είναι η ακτινοβολία. Δεν είναι δεν θα έπρεπε να πάρουμε αυτό το δρόμο ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε εμείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω μιλήσει με αεροπορικές εταιρείες που φοβούνται ε, ακόμη και περισσότερες μεγαλύτερες ουρές ε, στα αεροδρόμια επειδή θα φοβούνται οι επιβάτες να περάσουν από σαρωτές, από μηχανήματα που δεν θεωρούν ότι είναι ασφαλή. Ναι, είναι σαφές ότι ορισμένα μηχανήματα δεν είναι ε, εντάξει, όπως για παράδειγμα αυτές που ανέφερα στο Μάντσεστερ και στο Χίθρο και κάνουν και κάποιο είδους προφάιλινγκ, άλλωστε στα αεροδρόμια αυτά μέσω των μηχανημάτων και εγώ διαφωνώ καθέτος η κυρία Στύπο είπε ότι η ασφάλεια δεν μπορεί να σαρωθεί, συμφωνώ απολύτω, και η κυρία Μποσκούρτ με ρώτησε για τις ελάχιστες προδιαγραφές. Αν δείτε ε, την αρχική μου έκθεση, εμείς διατυπώσαμε τις ελάχιστες προδιαγραφές και ο κύριος Γκράντες, ο κύριος Δεγκράντες, ε, ε, ε, επίσης αποσαφήνισε τα πράγματα και σε μένα μου είπε το βασικότερο πράγμα είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα, το να είναι εθελοντικό και η προστασία δεδομένων δεν ε, είναι ο τρόπος να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι σε αυτό το τμήμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων μπορούμε να συμφωνήσουμε. Για να δω τι άλλο δεν απάντησα. Τους κανόνες γύρω από τους αρωτές, ναι. Θα ήθελα να το θέσω και αυτό. Ένας αρωτής μπορεί να είναι τέλειος, κάλιστος και νομίζω ότι έχω δει σαρωτές που είναι των προδιαγραφών που θα επιθυμούσαμε εμείς. Όμως είναι πολύ σημαντικό επίσης να μην επιλέγουμε ε, ποιοι επιβάτες θα περάσουν από το σαρωτή και ποιοι όχι ε, και πρέπει αυτοί που χρησιμοποιούν τους σαρωτές να καταρτίζονται ορθά, ώστε αν κάποιος περάσει από το σαρωτή και θεωρείται ότι δεν είναι επικίνδυνος, να μην γίνεται μετά προφάιλινγκ του ανθρώπου αυτού. Έχω και κάτι ακόμη που θα ήθελα να προσθέσω. Είπε ο κύριος Ντεγκράντες ότι κρίμα είναι που δεν περιμέναμε την έκθεση αυτή για να μπορέσουμε να εγκρίνουμε και τη δικιά μας. Ναι, μα και εμείς θέλαμε να σας επηρεάσουμε στη δουλειά σας αλλά αν θέλετε να περιμένουμε την έκθεσή σας, νομίζω ότι θα έπρεπε η Επιτροπή σας να καθυστερήσει την ψηφοφορία της, γιατί διαφορετικά δεν, δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε στην δική σας έκθεση. Αυτή είναι η απάντησή μου στον κύριο Ντεγκράντες. Ελπίζω να μην ξέχασα τίποτα. Αυτά ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Αυτά ε, ήθελε να πει η κυρία Σαρτζεντίνη. Κύριε Ντεγκράντες, θέλετε να πάρετε το λόγο. Μετά όμως θα πρέπει να δώσουμε και το λόγο στην κυρία Σαρτζεντίνη για να έχει εκείνη τον τελικό λόγο. Λίγο σύντομα μόνο γιατί έχουμε καθυστερήσει. Ναι, ευχαριστώ βεβαίω. Η κυρία Σαρζαντίν είναι η κυρία τη έκθεση και εκείνη θα πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο. Δεν ε, έχω πρόθεση παραπάνω να βοηθήσω. Και θα ήθελα να πω ότι δεν διατύπωσα κατηγορίε κατά κανενός, Απλώ είπα ότι κάπως έτσι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη διαδικασία. Και μίλησα και με την κυρία Σαρζεντινή, Δικατηδίαν καθώς θεωρώ ότι θα πρέπει η Επιτροπή σας να έχει προφορικά έστω τις, ε, τα στοιχεία για την ουσία της εκθεσής μου. Η εκθεσή μου είναι ήδη διαθέσιμη στα Ισπανικά. Θα προχωρήσει τώρα στη μετάφραση. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες. Και θα δείτε, πιστεύω, ότι το σύνολο σχεδόν των ιδεών, των ανησυχιών που καταγράφονται, σας ε, καλύπτουν. Αντικατοπτρίζονται όλες οι ιδέες και οι ανησυχίες που εκφράστηκαν εδώ. Και θα ήθελα να αποφεύγουμε τους, τις δίκες προθέσεων, ε, Πρόεδρε. Η καταπαλέμηση της τρομοκρατίας απαιτεί να είμαστε πιο αποφασιστικοί Τα κράτη-μέλη έχουν καθήκον να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της τρομοκρατίας. Τα υφιστάμενα συστήματα δεν είναι ικανοποιητικά 100%. Και προκειμένου να τα βελτιώσουν, οι δημοσιαρχές οφείλουν να λάβουν τις βέλτιστες κατά την άποψή τους διτάξεις. Αλλά και αυτό δεν μπορεί να γίνει πάση θυσία, με κάθε τίμημα δηλαδή. Βεβαίως έχουμε το καθήκον της του πολίτη, αλλά όχι με κάθε τίμημα γιατί ε, δεν είναι αποδεκτό ας πούμε, το να θυσιαστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε. Χρειαζόμαστε μέσα προστασίας, που είναι πιο ε, εύστοχη νομίζω διατύπωση από το να μιλούμε για μέτρα ασφαλείας. Άρα χρειάζεται μια λύση η οποία να επιτρέπει να βελτιωθούν τα υφιστάμενα συστήματα, μια λύση η οποία να εξασφαλίζει και την ε, τήρηση αρχής αναλογικότητας μεταξύ των ε, υφισταμένων συστημάτων και να προσφέρει βέβαια την απαραίτητη προσθέμενη αξία, σεβόμενη ωστόσο και τις ε, θεμελιώδεις, θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα. Όλα όσα λέτε λοιπόν εσείς εδώ τα έχω ήδη υπόψη και περιγράψει στην έκθεσή μου. Ίσως θέλετε να τροποποιήσετε το χρονοδιάγραμμα. Αυτό δεν είναι θέμα δικής μου αρμοδιότητας. και νομίζω ότι η γνωμοδότησή μου αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες της Επιτροπής των Πολιτικών Ελευθεριών κατά ικανοποιητικό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε την έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δύο πράγματα έχω να συμπληρώσω για να δώσω απάντηση. Μια παρατήρηση καταρχά τη κυρία Σνετφέλντο προ το τι είναι αυτό το οποίο επιδιώκουμε και τι εξετάζει ο, ο σαρωτής μέσα ή έξω. Έχετε πολύ σωστό, είναι πολύ εύστοχη η παρατήρηση σας. Εάν πρόκειται για υλικό κρυμμένο με συγκυλότητες του σώματος, αυτός ο σώματος δεν είναι χρήσιμος. Μόνο οι ακτίνες χ μπορούν να, να διαγνώσουν κάτι τέτοιο. Και δεύτερον, το εμπορικό συμφέρον. Από ό,τι βλέπω και από ό,τι ακούω, υπάρχουν μεγάλα εμπορικά συμφέροντα. Αυτά λένε και οι εμπορικές εταιρείες οι οποία διαδίδουν διαφορετικές πληροφορίες για το τι είναι ασφαλές, τι δεν είναι, ποιο σύστημα είναι αποτελεσματικό και ποιο δεν είναι. Και ως εκ τούτου καταλήγω και πάλι στο συμπέρασμα που τίνει προς τις ακτίνες Χ. Δηλαδή ε, το εμπορικό συμφέρον είναι αυτό το οποίο προσπαθεί να διατηρήσει στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων το θέμα των ακτίνων Χ, προκειμένου να κερδίσουν χρήματα. Εν τέλει, 16 Μαρτίου προβλέπεται η ψηφοφορία. Την επόμενη Παρασκευή έχουμε την προθεσμία για την καταστροπολογία. Στο 12 το μεσημέρι. Ήθιστε πρώτα να ψηφίσετε μια χρονομοδότηση και μετά η κυρία έκθεση. Εάν επιμένει ο κύριος Δεγραντεγράντες να λάβουμε υπόψη την έκθεσή του και εκτιμώ την πρόθεσή του, θα πρέπει να καθυστερήσουμε τη δική μας διαδικασία, αλλά θα πρέπει και εκείνος να καθυστερήσει τη δική του διαδικασία αντίστοιχα. Αντίρρηση δεν έχω εγώ ως προς τη δική μας την πλευρά, αλλά θα πρέπει και η Επιτροπή των Μεταφορών να αναβάλει τις σχετικές διαδικασίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σαρσεντίνη. Για να ολοκληρώσουμε τώρα τη συζήτηση. Τροπολογίες θα πρέπει να καταθέσουμε μέχρι τις 4 Μαρτίου. Το μεσημέρι 12. για να γίνει ψηφοφορία όπως προβλέπετε. Ευχαριστώ για τη συζήτηση και πάω στο επόμενο θέμα, το υπαριθμόν 15. Sorry, I that. Κύριε Σαρζεντίνη, υπάρχει κάτι το οποίο ίσως δεν κατάλαβα, Πρόεδρε. Ναι, είπα τροπολογίες 4 Μαρτίου. Έχετε αντίρρηση. Θέλετε αναβολή. Δεν άκουσα τον κύριο Ντεγκράντε, δεν μα είπε ότι πρόκειται να αναβάλει τη δική του τη διαδικασία, άρα δεν μπορούμε εμείς να, να αναβάλουμε τη δική μας, άρα όχι. Κύριε Ντεγκράντε, όχι δεν είναι ότι δεν το θέλω, είναι ότι δεν, δεν περνάει το χέρι μου. Οι διαδικασίε έτσι έχουν. Εγώ, Φερρυπίν, θα είμαι συντάκτη γνωμοδότηση σε μια υπόθεση που έχει την ε, κατ' ουσίαν έκθεση η Επιτροπή σα στην Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων για την Καταπολέμηση τη Δημοκρατία και δεν θα γνωρίζω καν το περιεχόμενο τη έκθεση. Κυρία Σαρζεντινή, ναι, μα εσεί είστε ο αρμόδιο κατ' ουσίαν αυτή τη στιγμή. Στο χέρι σα είναι. Εμεί πρέπει να είμαστε έτοιμοι απολώ πριν από τη δική σα ψηφοφορία. Καλό θα ήταν να έχουμε το κείμενο αφού δούμε την έκθεσή σας. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο που δεν τον βλέπουμε τώρα. Εγώ είμαι τώρα στη δική σας διάθεση. Κύριε Στεκράντος. Πρόεδρε, δεν βλέπω καμιά αντίρρηση, αλλά δεν περνάει από το χέρι μου. Είναι θέμα αρμοδιότητα, είναι θέμα μάλλον απόφαση Επιτροπή των Μεταφορών. Να του το προτείνω εγώ, αν δεν υπάρχει αντίρρηση. 15 Μαρτίου εγώ καταθέτω την έκθεσή μου. Άρα Μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Στον κύριο Σίμψον, λοιπόν, τον πρόεδρο τη Επιτροπή των Μεταφορών, θα ζητήσω, θα μεταφέρω μάλλον ότι η Επιτροπή των Μεταφορών ζητεί μια παράταση των σχετικών ε, προθεσμιών. Αν δεν έχετε αντίρρηση, πολύ ευχαριστώ. Κύριε Σαρζαντίνη, σα διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση από πλευρά μου ω προ την παράταση των ε, προθεσμιών. Ο πρόεδρο. Καλώς με την προοπτική ότι θα συντονίσουμε τις ημερομηνίε μας προχωρούμε. Εμείς προς το παρόν διατηρούμε 4 Μαρτίου την προθεσμία για και βλέπουμε. Επιφυλασσόμενοι όπως είπα ότι μπορεί να συντονίσουμε τελικά τις προθεσμίες αυτές με την Επιτροπή των Μεταφορών. Και πάμε τώρα στο σημείο 15. Συντονιστές έχουμε μετά. Τώρα έχουμε το 15. Στρατηγική ασφάλειας. Την έχουμε προβλέψει για περίπου μισή ώρα και μετά θα γίνουν οι συνεδρίε των συντονιστών. Έχετε καμιά αντίρρηση, κυρία Πουσούτιλ. Πρόεδρε, έχουμε πολλά για του συντονιστέ. Προφανώ δεν έχουμε χρόνο να δούμε και το 15. Μέσα σε 5 λεπτά δεν προλαβαίνουμε ούτω ή άλλω. Είναι ντροπή να το κάνουμε έτσι. Επομένω πρέπει να αποφασίσουμε, θα κάνουμε συνεδρίε των συντονιστών ή όχι. Δεν έχει γίνει συνεδρίε των συντονιστών εδώ και τρει εβδομάδε. Και πολλέ είναι οι εκκρεμίε αποφάσει. Βεβαίω και θα γίνει συνεδρίε των συντονιστών, λέει ο πρόεδρο. Το θέμα είναι μήπως, να μην κάνουμε το 15. Η κυρία Μπορσελίνο είναι εδώ η συγκεκριά. Μπορούμε να ξαναδούμε το πρόγραμμα. Αλλά πρέπει να συμφωνήσουν οι πολιτικές ομάδες. Γιατί διαφορετικά είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε την μέρη διάταξη. Κύριος Μωράς. Η κυρία Πορσελίνη, η οποία περιμένει τόση ώρα για να παρουσιάσει την εκθέση της. Ίσως να τη ρωτήσουμε αν προτιμάει τώρα να το παρουσιάσει πολύ σύντομα ή αλλιώ να τη δώσουμε πιο πολύ χρόνο σε μια άλλη συνεδρίαση γιατί περιμένει εδώ και ώρα. Και είναι σημαντικό βέβαια θέμα αυτό τη ιστορική στρατηγική στρατηγικής, Κυρία Προσελίνη. Εγώ είμαι στη διάθεσή σα να περιμένω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα ε, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Τώρα να το κάνουμε έτσι στα βιαστικά ε, μέσα σε πέντε λεπτά γιατί έχετε άλλες δουλειές μετά δεν μου φαίνεται ότι είναι σωστό. Πρόεδρος. Άρα θα είχατε την ευγενή καλοσύνη να δεχτείτε να αναβάλουμε το θέμα αυτό για την επόμενη συνεδρία Δεν πρόκειται για ευγένεια. Δεν, έχουμε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, λέει η κυρία Μπορσελίνο. Δεν είναι ένα θέμα που μπορεί να συζητηθεί έτσι στα βιαστικά μέσα σε πέντε λεπτά. Δεν το νομίζω. Εντάξει, λέει ο Πρόεδρος, αν συμφωνείτε κι εσείς ε, θα αναβάλουμε το θέμα αυτό για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας, ούτως ώστε τώρα να προχωρήσουμε στη συνεδρίαση ε, ε, των συντονιστών που έχει πολύ φορτωμένη ημερήσια διάταξη. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε, μπορείτε να ζητήσετε από τη Γραμματεία να φροντίσει ώστε το θέμα της κυρίας Μπορσελίνου να ξαναμπεί ε, την κατάλληλη χρονική στιγμή και πάλι στην ημερήσια διάταξη. Βεβαίως, βεβαίως, οπωσδήποτε. Θα έχουμε σίγουρα το θέμα της κυρίας Μπορσελίνου. Θα το έχουμε υπόψη μας. Ωραία, τώρα ε, συνάντηση των συντονιστών και κλεισμένων των θυρών. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας στις συζητήσεις που είχαμε. Ευχαριστούμε και όλους τους παρευρισκόμενους ε, και τους παρακαλούμε να μας ε, αφήσουν να προχωρήσουμε στη συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών ε, για την συνάντηση των συντονιστών.